Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη που σας άφησα να περιμένετε λίγο. Ε, ε, είχα μια άλλη υποχρέωση και γι' αυτό άργησα. Εν πάση περιπτώσει, ας αρχίσουμε τώρα τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ήτρε. Έχουμε συνεδρίαση σήμερα το πρωί, ε, σήμερα το απόγευμα ακρόαση και την Πέμπτη το πρωί. Ε, Ξεκινάμε με την υιοθέτηση της ημερήσιας διάταξης, εάν δεν έχετε σχόλια, να θεωρήσουμε πως εγκρίνεται. Χωρίς αλλαγές, δεν βλέπω να υπάρχουν σχόλια. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Δεν έχω τίποτα ιδιαίτερο. Θα σας ζητήσω να ε, τηρήσουμε ενός λεπτοσυγή, αλλά ε, λίγο πριν την ψηφοφορία, όταν θα έχουν έρθει και άλλοι συνάδελφοι. Γιατί είναι η πρώτη επέτειος των τρομοκρατικών επιθέσεων ε, στην πόλη μας, στις Βρυξέλλες όπου εμείς εργαζόμαστε, ζούμε τρεις-τέσσερις μέρες την εβδομάδα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε την αλληλεγγύη μας, να συμπαρασταθούμε στα οικογένειες των θυμάτων. Και αλληλεγγύη μεταξύ μας επίσης είναι πολύ σημαντική. Πρόταση τώρα είναι το επόμενο σημείο, το 3 ε, για τη χρήση γης, αλλαγές της ε, γης, τη δασοκομεία, στο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια. Με ορίζονται το 2030. Πρόκειται για ένα τροποποιητικό κανονισμό προηγούμενου, το του προηγούμενου κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Και η συγκήτριά μας, η Μαρίζα Ματία, σήμερα αντικαθίσταται από τον κύριο Χαβιέρ Μπενίτο Σιλουάγκα και θα εξετάσουμε λοιπόν ε, το σχέδιο γνωμοδότησης που αφορά την χρήση της γης, τις αλλαγές στη χρήση της γης και τη δασοκομεία που αποκαλείται και λούλουσι η επί αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Εμείς θα συντάξουμε γνωμοδότηση. Η πρόταση στόχο έχει να περιορίσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από την χρήση της γης και τη δασοκομεία, ενθαρρύνοντας ας πούμε την ε, βιώσιμη δασοκομεία και ε, πρόκειται για συνέχιση των στόχων μετά την εκπνοή του Κιώτο το 2021. Η πρόταση Λουλουσιέφ είναι πολύ, ε, πολύ ε, σημαντική για την Επιτροπή μας γιατί αγγίζει πολλά ζητήματα που εμπίπτουν στις δικές μας αρμοδιότητες όπως η έρευνα, η καινοτομία, η παρακολούθηση, εποπτεία της χρήσης γης με δορυφόρους αλλά αφορά και την βιομηχανική μας πολιτική που βασίζεται στην δασοκομεία. δηλαδή το τμήμα της βιομηχανίας που βασίζεται στη δασοκομεία. Χαβιέρ Μπενίτο Ζιλουάγα, στη θέση της Μαρίζα Ματίας. Από την ΚΟΥ έχετε το λόγο. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όντως η σύντροφος Μαρίζα Ματίας δεν, μπορούσε να είναι παρούσα σήμερα και ζητά συγγνώμη, αλλά ταυτόχρονα βρίσκεται σε μια αποστολή παρακολούθηση των εκλογών στο Ανατολικό Τιμόρ και ε, γι' αυτό και δεν ήταν δυνατό να είναι σήμερα παρούσα. Αλλά θα σας εκθέσω εγώ κάποιες ιδέες που μου ε, μεταβίβασε για την σύνταξη αυτής της γνωμοδότησης. Καταρχάς, η συγκήτρια πιστεύει πως αυτή η γνωμοδότηση θα είναι σημαντική για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να... Ε, ανταποκριθεί στους στόχους ε, της Συμφωνίας του Παρισιού με ικανοποιητικό τρόπο τόσο από την περιβαλλοντική άποψη όσο και από την οικονομική και κοινωνική και ότι επιπλέον λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές καταστάσεις, πλαίσια και μοντέλα διαχείρισης που υπάρχουν ε, στα διάφορα κράτη-μέλη. Κατά δεύτερο λόγο, η συγκήτρια θεωρεί πως η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ένα σημείο εκκίνησης εξαιρετικό για, την, για εργασία και ακριβώς ε, αγγίζει σημεία κλειδιά μεταξύ των οποίων τα εξή για τη δική μας Επιτροπή, αύξηση των κονδυλίων για την έρευνα και την ανάπτυξη, για τη διαχείριση των δασών, δεύτερον η χρήση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων παρατήρησης με μεσοδορυφόρου, όπως το Κοπέρνικος, για να παρακολουθούμε την ανάπτυξη και της χρήσης της γης έπειτα για την διαφοροποίηση την διατροφική και ε, ε, επίσης αλλάζουν η νομική βεβαιότητα για τους ε, φορείς, τους ιδιωτικούς αλλά και για τα κράτη. Βελτιστοποίηση δε του συστήματος παρακολούθησης και εποπτείας τόσο σε κρατικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με συγκεκριμένες αναφορές για κάθε τομέα και έκτον ένα σύστημα, να στοχεύσουμε μάλλον σε ένα σύστημα διαχείρισης της γης ε, σε ε, σύμμορφο προς τις αρχές της οικονομίας ε, της κυκλικής. Τέλος, θεωρεί σημαντικό ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε ευρία συνένεση όσο γίνεται ανάμεσα σε όλες τις ομάδες για αυτή την έκθεση και γι' αυτό και είμαστε ευτυχείς που μπορέσαμε να λάβουμε αυτές τις προτάσεις και έτσι να μπορέσουμε να συμβάλλουμε όλοι στο να συνταχθεί ένα όσο γίνεται καλύτερο κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφε, και θα ακούσουμε τώρα τους Σκιώδης. Η κυρία Γιούσο από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πόσο χρόνο μου δίνετε? Δύο λεπτά, δύο λεπτά έχετε. Αντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ε, ναι, θα προσαρμοστώ στα δύο λεπτά. Αυτή η πρόταση, όπως σωστά είπε ο ο εκπρόσωπος της εισηγήτριας θεσπίζει κάποιες ε, περιόδους ε, εφαρμογής, ε, υλοποίησης αλλά και μορφές καταμέτρησης που κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά περίπλοκη αλλά και μια σειρά από ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε την περίοδο 2021-2025 αλλά και το 2026 μέχρι 2030, αλλά δεν λέει τίποτα για ευελιξίες για την ε, ε, ε, μετέπειτα περίοδο και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Τώρα, συγκεκριμένη καταμέτρηση για προϊόντα ξύλου είναι εξαιρετικά περίπλοκο το σύστημα που προτείνεται εδώ αφήνει πολύ χώρο στην υποκειμενικότητα για να γίνουν οι μετρήσεις και οι υπολογισμοί. Επίσης υπάρχει ένα στοιχείο καταμέτρησης των φυσικών ε, καταστροφών ή των θεομηνιών που εξαιρεί τις χώρες από την καταμέτρηση σε περίπτωση που χτυπήσουν τέτοια φαινόμενα. Λοιπόν, να μείνω στα όσα είπε η, η Η βιοπικιλότητα, όπως το λέει και η συγγήτρια, ε, θα πρέπει και η προστασία αυτής ε, θα πρέπει να είναι συνεπής με την, ε, σε πολιτι... σχετικές πολιτικές και θα πρέπει να μπορούν να πιστοποιηθούν όλα αυτά όπως το προτείνει στην τροπολογία της 10. Ε, έχουμε και τις περιοχές Natura 2000, θα πρέπει να πιστοποιηθούν για να μπορέσουμε, λέει, να τις καταμετρήσουμε. Αυτό νομίζω πως είναι υπερβολικό. Ποιος θα το κάνει όλη αυτή τη δουλειά χρειάζεται περίοδος προσαρμογής και όσον αφορά την ε, ε, ε, δορυφορική παρακολούθηση θα πρέπει επίσης να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος. Η, συγκήτρια προτείνει σχέδιο δράσης για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις ε, σχετικές ενέργειες από το 2040 και μέχρι και το 2070. Αλλά πιστεύω εγώ πως είναι πολύ μακροπρόθεσμα όλα αυτά. Ε, δηλαδή ε, τέτοιο είδους προγράμματα και σχέδια δεν μπορούν να τα ετοιμάσουν όλα τα κράτη. Ο πρόεδρος διακόπτει. Ναι, ένα δευτερόλεπτο. Όσον αφορά τώρα τη σύγκριση των στοιχείων ανάμεσα στα κράτη-μέλη, ναι, πρέπει να σας τα πω. Πρέπει να σταματήσω. Ε, κοιτάξτε, μιλήσατε τρία λεπτά, όχι δύο που σας είπα. Λυπούμε. Άντε, μία-δύο φράσεις για να τελειώσετε Τώρα, για τις μεταφορές ανάμεσα στα κρατημέλη δεν νομίζω πως υπάρχει κάποια βάση για να δικαιολογεί αυτή την ευελιξία του 25%. καλύτερα θα ήταν να μείνει στο 5%. Και θα πρέπει το κάθε κράτος μέρος να μπορεί να χρησιμοποιήσει όποτε το επιθυμεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κομπούλα Νάτρη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να περιοριστώ στο, στα ζητήματα τα οποία είναι τα πιο σημαντικά για την Επιτροπή μας ε, Καινοτομίας Ενέργειας και Έρευνας. Πρέπει λοιπόν εμείς ε, να ασχοληθούμε με αυτά περισσότερο, γιατί η ΕΝΒΗ θα εξετάσει πιο πολύ τα περιβαλλοντικά. Εμά λοιπόν μας ενδιαφέρει περισσότερο η βιοοικονομία και γι' αυτό θα καταθέσω τροπολογία σε ό,τι αφορά τα προϊόντα ξυλία να αποτελέσουν ξεχωριστή κατηγορία για να δούμε τι δυνατότητα υπάρχει. Μπορούμε να εξετάσουμε και την βιώσιμη αντικατάσταση ε, προϊόντων ε, των ορικών, ορικών καυσίμων και γενικότερα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα βιώσιμο ε, δοσοκομικό μοντέλο σε πολλές χώρες, ε, αλλά να αξιοποιήσουμε και τέτοια μέσα σε χώρες που δεν το έχουν πράξει στο παρελθόν. Δεν θα πρέπει λοιπόν να ε, κόβουμε δέντρα για να φτιάξουμε σπίτια, αλλά θα πρέπει να τα όλα αυτά υπόψη ε, και στην οικονομική δραστηριότητα. Κάποιε χώρε χρειάζονται περισσότερη ε, χώρα. Πρέπει λοιπόν να φυτέψουν νέα δάση. Όμω υπάρχουν χώρε που ήδη καλύπτουν κατά 75% από δάση. Επομένω είναι λίγο περιοριστικό να λέμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα καλύτερο όταν κόβουμε ένα δέντρο πρέπει να φυτεύουμε και ένα δέντρο. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια διαχείριση δοσοκομική και από εδώ και πέρα. Για τα επίπεδα αναφορά είναι πολύ δύσκολα γιατί ε, άλλε χώρε αξιοποιούν το 85% των δασών ανα πάσα στιγμή, ενώ άλλε 40%. Πρέπει λοιπόν να είναι βιώσιμο το μέλλον και η διαχείριση των δασών να ε, είναι τέτοια που να μα επιτρέψει να συνεχίσουμε με καλύτερο τρόπο για τα δεδομένα, κοπέρνικους και ούτω καθεξής. Ε, μπορούμε να εργαστούμε από κοινού και για λόγους διαφάνειας πρέπει να διαμορφωθεί ένα καλό πρότυπο και για το μέλλον της δοσοκομείας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φέντερλε από τους Φιλελεύθερους. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την έκθεση. Είναι μια καλή βάση για τη συνέχιση των συζητήσεων. Ο ίδιος ο φάκελος βέβαια είναι σημαντικό τμήμα ε, της δέσμης ε, για την, κλιματική αλλαγή Και σε ένα πρόσφατο πάλι αναφέρεται ότι η διατήρηση ενίσχυση των συγκεκριμένων πόρων ε, διατηρώντας ε, ε, και την ξυλία και το καθεξής από το δάσος θα μας δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα. Συμφωνώ εδώ ότι οι υπολογισμοί και τα επίπεδα αναφοράς θα είναι το κέριο ζήτημα. τα δάση δεχάνουν διαφορετική διαχείριση ε, σε διάφορα σημεία τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρουμε ότι υπάρχουν και διαφορετικοί τύποι ε, δασών. Σε άλλε χώρε έχουμε μικρού ιδιοκτήτε των δασών, ενώ αλλού είναι κρατικά. Δημόσια. Έχουμε και ένα σύστημα που υλοποιήθηκε, εγκρίθηκε υπό το Κιώτο και έχει οδηγήσει σε αύξηση των δασών εδώ και έναν αιώνα σχεδόν συνεχώς θα ήθελα σε μια τροπολογία να προτείνω υπολογισμούς βάσει του ειδικού μοντέλου που είναι πραγματικά βιώσιμο, διασφαλίζει αύξηση της βιομάζας, αλλά διασφαλίζει και ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα προϊόντα που προκύπτουν από το δάσος και για την καταπολέμηση ε, της κλιματικής αλλαγής. Έχουμε την εντύπωση ότι με τα επίπεδα αναφοράς που προβλέπονται τώρα πρέπει να υπάρχει 9% αύξηση κάθε χρόνο. Όμως ε, τελικά θα έχουμε μόνο ε, δάση στη Σουηδία. Θα πρέπει να ε, καταργήσουμε γεωργικές εκμεταλλεύσεις για να φυτέψουμε δέντρα. Ε, πρέπει να συσχετίσουμε και την ζήτηση των δασικών προϊόντων με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικονομία. Μπορεί να υπάρχουν και φυσικές αιτίε όπως ε, πυρκαγιές ε, και ούτω καθεξής. Θα επανέλθουμε λοιπόν με συγκεκριμένε προτάσεις γιατί θεωρούμε ότι η Ήτρε μπορεί να συμβάλλει σημαντικά σε αυτή τη συζήτηση που γίνεται στην Ένδη και στην Άγκρη. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Γιάβορ από τους Πράσινους. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεσης που αποτελεί καλή βάση συζήτησης. Μερικές παρατηρήσεις για ζητήματα που εν μέρει έχουν ήδη θυγεί. Πρώτον, βέβαια ο κανονισμός ε, Λουλουσιέφ είναι σημαντικός, όμως αποτελεί ένα στοιχείο μιας ευρύτερης δέσμης ε, που άπτεται του κλίματος. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχουμε κατά νου και τις υπόλοιπες ε, προτάσεις. Μεταξύ άλλων και την πρόταση ESR. Να λάβουμε υπόψη τις μακροπρόθεσμες ε, Δεσμεύσει ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την απαλλαγή από τον άνθρακα, τις ε, υποσχέσεις ε, στο πλαίσιο της συμφωνία των Παρισίων. Θα πρέπει λοιπόν και η Λουλουσιέφ να ενταχθεί στο πλαίσιο αυτών των μακροπρόθεσμων στόχων. Νομίζω ότι είναι σημαντική και η στόχη της βιοπικιλότητας, γιατί αναπόφευκτα θα πρέπει να, υπο... να ληφθεί και αυτά υπόψη. Επόμενο είναι οι λογιστικοί κανόνες. Νομίζω ότι επιτέλους θα πρέπει να εξετάσουμε όλα αυτά τα στοιχεία σε αυτό το πλαίσιο. Γι' αυτό προτείνω ένα συγκεκριμένο λογιστικό σύστημα και πρέπει να συμπεριλάβουμε και τους υγροβιότυπους και τους τριφώνες ε, ε, σε αυτό το πλαίσιο για να έχουμε ένα διαφανές και ακριβές λογιστικό σύστημα. Το ζήτημα της ευελιξίας με τον κανονισμό ESR πρέπει να τεθεί επιτάπητος για να δούμε ποια είναι τα αποδεκτά επίπεδα του μηχανισμού ευελιξίας. Και κατά τελευταίο, έρευνα και ανάπτυξη που είναι σαφώς ε, το πλέον σημαντικό για την Επιτροπή Ήτρε. Είδαμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε, στις Ηνωμένε Πολιτείε, η έρευνα και ανάπτυξη που συνδέεται με το κλίμα θα χρηματοδοτηθεί στο μέλλον και νομίζω ότι και η Ευρώπη τώρα έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει τον ηγετικό ρόλο σε ό,τι αφορά την έρευνα και ανάπτυξη, όμως απαιτείται πραγματική αφοσίωση και χρηματοδότηση από ευρωπαϊκής πλευράς, αλλιώς η Κίνα θα αναλάβει τον ρόλο. Ας αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα λάβει το λόγο η κυρία Σάιμον Κέι από τη Γενική Διεύθυνση Climate. Ο κύριος Κέι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν πειράζει που κάνατε λάθος. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να έρθω εδώ, να ακούσω την ανταλλαγή απόψεων. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον Άκουσα τις απόψεις της Επιτροπής Ήτρε για το θέμα αυτό, το οποίο φυσικά ε, συζητιέται και σε γενικότερο πλαίσιο, σε συνδυασμό με τις άλλες σχετικές προτάσεις. Θα θέλαμε πράγματι να διασφαλίσουμε πως υπάρχει ε, κατανόηση για το ότι το πακέτο αυτό, οι δέσμοι μέτρων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορεί να ανταπεξέλθει στι ανησυχίες που έχει εκφράσει και το Συμβούλιο και οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς κατά τη διάρκεια της ε, διαβούλευση και να ταιριάζουν όλα τα μέτρα ε, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ε, αποτελεσματικό πακέτο το οποίο θα αντιμετωπίσει γρήγορα τις προκλήσεις που υπάρχουν. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για την έρευνα και την ανάπτυξη και για το Γαλιλαίο και για όλες τις προτάσεις που αναφέρονται στο σχέδιο έκθεσης. Αυτά φυσικά τα έχουμε κοιτάξει και εμείς και τα έχουμε συμπεριλάβει στις προτάσεις μας υπό το εφιστάμενο πλαίσιο του Λουλουσιέφ, αλλά επίσης είναι και ένα θέμα το οποίο να γνωρίζουμε ε, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και φυσικά υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες οι οποίες ε, έχουν συμμετοχή στο νομοθετικό αυτό έργο. Πρέπει να προσέξουμε οι προτάσεις να είναι ε, καλές, να επικαιροποιηθούν οι φυστάμενοι κανόνες, έτσι ώστε να συμφωνούν το πρώτο μέρος της Συμφωνίας των Παρισίων και ε, αυτό νομίζω πως θα πρέπει να είναι το κύριο μέλημά μας. και μετά μπορούμε να δούμε τα ωφέλη και ποιους τομείς ε, θα ε, αφορούν. Σας ευχαριστώ πολύ. want to say... Ευχαριστώ. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι. Ε, θέλω μόνο να ευχαριστήσω τους Κιώδης για τις ε, ενδιαφέρουσες απόψεις τους και εγώ φυσικά θα διαβιβάσω στην εισηγήτρια όλες αυτές τις σκέψεις και προβληματισμούς. Ε, να επαναλάβω ότι η ε, ελπίδα μας είναι να έχουμε μεγάλη συνένεση και μια καλή έκθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών 25 Μαρτίου. 27 Μαρτίου το μεσημέρι, ψηφίζουμε 11 Μαΐου 2007, 27 λοιπόν Μαρτίου, προθεσμία για τροπολογίες. Στις 12 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή, παρότι λείπει, αλλά ευχαριστώ πολύ και τους κοιόδες εισηγητές και όλους εσάς ε, συμπεριλαμβανομένες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά είναι το επόμενο θέμα μας. Η συγητής είναι ο κύριο Κρασνοντεύσκη. Κατόπιν δημοσίευσης της ε, πρότασης κανονισμού το Σεπτέμβριο του 2016, τα πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά ε, είναι το θέμα, είναι ο ίδιος ε, τίτλο με την νομοδότησή μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις και όραμα έτσι ώστε να επικαιροποιηθούν οι φυστάμενοι να επικαιροποιηθεί η φυστάμενη νομοθεσία. Ένας γενικότερος τίτλος, στόχος είναι να μειωθούν ε, οι διαφορές και να εξομαλυνθεί η νομοθεσία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι επιτροπές Ήτρε, Ίμκο και Κάλτε ακολουθούν την ε, καθήλυνα αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τον κανόνα 53 και ο συνάδελφος κ. Κρασνοτέψκη έχει συντάξει το σχέδιο γνωμοδότησης και θα του δώσω αμέσω το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Αυτή η πρόταση οδηγίας πράγματι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για πολλούς. Δεν περίμενα να είναι τόσο σημαντικό το θέμα για τόσο πολλούς διαφορετικούς φορείς. πρόταση αυτή ενδιαφέρει μια πληθώρα ομάδων από συγγραφείς, εκδότες, ε, όσοι ασχολούνται με το χώρο του κινηματογράφου, του θεάματος γενικότερα, αλλά και ε, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του διαδικτύου. Και πέρα από ορισμένα δύσκολα ζητήματα, υπάρχει γενικά μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα. Εδώ υπάρχουν τέσσερις ε, επιτροπές ε, που ασχολούνται με το θέμα αυτό, οπότε υπάρχει ένας ε, κάποιος ανταγωνισμός. Εγώ προσπάθησα να είμαι λιτός και στη γνωμοδότησή μου, μετά φυσικά από διαβούλευση με τη γραμματεία της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, προσπάθησα να εστιάσω σε θέματα τα οποία είναι οι κύριες αρμοδιότητες της δική μας επιτροπής, δηλαδή ε, το data mining. Γνωρίζω πως ε, οι σκιώδες εισηγητές θέλουν να αναφερθούν με τις τροπολογίες τους και σε άλλα θέματα, αλλά σας παρακαλώ να μην ξεχνάμε ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Επιτροπής μας. Τα άρθρα όπως το 11 και το 13 είναι ε, δύσκολη περίπτωση, είναι αρκετά αμφιλεγόμενα και υπάρχει ενδεχομένως μια σύγκρουση αρμοδιοτήτων. Η δική μου προσέγγιση ήταν πιο ελεύθερη. Συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ύπαρξη ενός υποχρεωτικού καταλόγου που θα αφορά τη χρήση ε, των ε, δεδομένων αυτών που ε, συλλέγονται που είναι αποτέλεσμα αυτή τη εξόριξη δεδομένων. Εγώ πιστεύω πω ε, κάποιε ομάδε θα πρέπει να έχουν ε, άδεια χρήση. Για παράδειγμα, διάφοροι επιστημονικοί οργανισμοί, διότι πρέπει να ακολουθήσουμε τις ε, τεχνολογικές εξελίξεις και ας μην ξεχνάμε πως υπάρχουν και αρκετές εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με την επιστημονική έρευνα. Αυτή η διάκριση λοιπόν ανάμεσα σε εμπορικές και μη εμπορικές επιστημονικές δραστηριότητες νομίζω πως είναι κάπως επίπλαστη. Ακριβώς διότι τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας, ένα διδακτορικό για παράδειγμα, πολλές φορές ε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς και να έχουν οικονομικά ωφέλη. η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών είναι να συνδεθεί ακόμα περισσότερο η ε, επιστήμη με το εμπόριο. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως ε, εδώ κοιτάζουμε πολύ ε, συγκεκριμένα πράγματα. Πρέπει να διευρύνουμε λίγο τους ορίζοντές μας και να δώσουμε τη δυνατότητα πρόσβασης σε χρήστες οι οποίοι έχουν, έχουν κάποια νομική βάση νομικά δικαιώματα για να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα. Όταν, για παράδειγμα, μπορείς, αγοράζεις ένα βιβλίο, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ε, το παράρτημα που αναφέρει η βιβλιογραφία. Αυτό μπορούμε να το εφαρμόσουμε και στον ε, ψηφιακό τομέα. και επίσης στην Επιτροπή Πολιτισμού, ε, ορμόδιος εισηγητής, ε, παροτρύνει να γίνεται καταστροφή δεδομένων, κάτι το οποίο δεν θεωρώ πως ε, είναι σωστό. Μετά, σε ό,τι αφορά το λογισμικό, υπάρχει ένας μια πρόταση περιορισμού της χρήσης του λογισμικού από πολύ συγκεκριμένες ομάδες, επιστήμονες για παράδειγμα. Τα. Από μένα σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Νίμπλερ από το Έλκο και οδησηγήτρια. Σα ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον εισηγητή για τη γνωμοδότηση, για τη δουλειά που έκανε και για την ανταλλαγή απόψεων που επέτρεψε να γίνει μεταξύ εκείνου και των σκεδών. Το, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δέσμη μέτρων για την ψηφιακή αγορά και την πνευματική ιδιοκτησία είναι σίγουρα ένα από τα σημαντικότερα νομοθετικά ε, επιτεύγματα ε, για την ψηφιακή αγορά. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην εξέτασή της. Εγώ θεωρώ προσωπικά πως η πρόταση της Επιτροπής είναι πολύ ισορροπημένη. Υπάρχουν βέβαια πολλοί τομεί οι οποίοι χρειάζονται διευκρίνηση, χρειάζονται περισσότερη σαφήνεια, όμω σε γενικές γραμμές είναι μια αρκετά εξισορροπημένη πρόταση. Προσπαθεί να λάβει υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερους ε, ε, τομείς και τα συμφέροντα όσο το δυνατόν περισσότερων ε, φορέων. Ο εισηγητής στη γνωμοδότησή του έχει ακολουθήσει μία συγκεκριμένη μελοθοδολογία με την οποία συμφωνώ. Εδώ βέβαια κύριε Πρόεδρε θα περιοριστώ και εγώ με τις τροπολογίες μου στα θέματα που αφορούν την δική μας επιτροπή, δηλαδή την έρευνα και την ε, επιστημονική κοινότητα. Γι' αυτό ε, σε ό,τι αφορά την εξόρυξη δεδομένων και ε, κειμένου νομίζω πως πρέπει να υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί αλλά να προσαρμοστούμε και στην ε, ψηφιακή εποχή. Τώρα, φτάνω σε αυτό που ήθελα να πω. Νομίζω πως δεν μπορώ να συμφωνήσω με την πρόταση του εισηγητή η οποία αφορά τις εξαιρέσεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξόριξη δεδομένων. Ο εισηγητής προτείνει να ε, δοθεί πρόσβαση όχι μόνο σε ορισμένους επιστημονικούς οργανισμούς και ομάδες ε, που έχουν άμεσο ενδιαφέρον, αλλά και σε ε, συγκεκριμένα άτομα, ιδιώτες. Τώρα, αυτό δεν με βρίσκει σύμφωνη, δεν θεωρώ σωστό να υπάρχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα για ε, εμπορικούς και μη εμπορικούς σκοπούς. Το θέμα βέβαια είναι να δούμε τι έχουμε στη διάθεσή μας και ε, να μην θεωρούνται αυτά τα δεδομένα ότι διατίθενται δωρεάν. Υπάρχουν δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς και εκεί πρέπει να υπάρχει κάποιο ε, αντίτιμο οι πολλές εξαιρέσεις στην πρόσβαση ή στην χρήση κειμένου, μουσικής, ε, περιεχομένου που αφορά, ε, που έχει πνευματικά δικαιώματα, πρέπει να ε, επανεξεταστεί. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η πρόσβαση σε, αυτά, σε αυτό το περιεχόμενο θα διατίθεται μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς. Εγώ λοιπόν έχω διαφορετική άποψη από τον εισηγητή και η ομάδα μου φυσικά και πιστεύω πως ε, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν δυνατότητες δωρεάν πρόσβαση σε, αυτά τα δεδομένα. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν και θα σταματήσω εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βέρνερ τώρα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή. Θα μιλήσω εκ μέρους της ε, συναδέλφου κυρίας Κόφιν, η οποία δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα. Η Τερίσα θεωρεί ότι το κείμενο αυτό αποτελεί μια πραγματική ευκαιρία για ε, να λειτουργεί η ψηφιακή ενία αγορά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προ όφελο όλων των ε, δημιουργικών κλάδων. ήδη πω είναι η ραχοκοκαλιά της ψηφιακής μας του ψηφιακού πολιτισμού και η εξόριξη δεδομένων χρειάζεται να συνδεθεί με μια δίκαιη αποζημίωση για τους ε, δημιουργούς, τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και να χαρακτηρίζεται φυσικά από διαφάνεια. Θεωρεί ότι το ε, άρθρο 3 είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι και η εξόριξη δεδομένων και κειμένου πρέπει να χρησιμοποιείται για καλό σκοπό και να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα αυτά θα ε, χρησιμεύσουν ε, για την ε, τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο. Η συνεργασία είναι επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο η σχέδιση συγκίτρια τονίζει πως πρέπει να διασφαλιστεί. Μετά, το άρθρο 20 αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και σύμφωνα με αυτό όσοι τα χρησιμοποιούν πρέπει να πληρώνουν και ένα αντίτιμο γιατί αυτή, τη φορά, γιατί αυτή την εποχή υπάρχουν τεράστια κέρδη από τη δωρεάν χρήση περιεχομένου που έχει πνευματικά δικαιώματα. Χρειάζεται λοιπόν να προστατευθούν οι δημιουργοί των οποίων το περιεχόμενο χρησιμοποιείται χωρίς ε, την συγκατάθεσή τους και χωρίς αποζημίωση. Τώρα, σε ό,τι φορά τα άρθρα 14 έως 16, η ε, Τζέιζα θα θέλει ε, να διασφαλιστεί και εδώ ότι η παροχή πληροφοριών θα είναι ε, χαρακτηρισμένη από ακρίβεια και πως οι δημιουργοί θα αποζημιώνονται επαρκώς για το ε, έργο που χρησιμοποιείται, για το, το έργο τους που έχει πνευματικά δικαιώματα και θα εξαλειφθούν οι πρακτικές αθέμη του ανταγωνισμού. Αυτό σε όλους τους τομείς και στον ε, τομέα των ε, ψηφιακών έργων. Μετά, σε ό,τι αφορά το άρθρο 11, η συνάδελφος ζητά την ε, κατάλληλη αποζημίωση των δημοσιογράφων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ε, δημοσιογραφική ανεξαρτησία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ριβαζή τώρα έχει το λόγο εκ μέρους των Πρασίνων. She she's gone. Λείπει. Από την ΚΟΕ θα μιλήσει η κυρία Κορνιλιά Ένστ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα ε, να αρχίσω λέγοντας ότι ναι, δεν θεωρώ πως η πρόταση της Επιτροπής ε, με βρίσκει σύμφωνη. Μάλιστα, τολμώ να πω πως ντρέπομαι για αυτό που διάβασα, ντρέπομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έκανε μία τέτοια πρόταση. Το, τώρα, το σχέδιο γνωμοδότησης νομίζω πως δεν αλλάζει ουσιαστικά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και θέλω να ασκήσω κριτική σε αρκετά ε, πράγματα, αλλά σε ό,τι αφορά το σχέδιο γνωμοδότησης να πω ότι οι ε, άδειε χρήσης είναι ένα πολύ προβληματικό σημείο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάνει αρκετές προσπάθειες για να διασφαλίσει την ανεξαρτησία των ε, δεδομένων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις μεγάλες εταιρείες ε, και επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και τους ε, μεγάλους ομίλους. Εμείς θεωρούμε πως η διατύπωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι λανθασμένη. Υπάρχει πολύ περιοριστική διατύπωση. Τα... Η χρονική περίοδος των 25 ετών που προτείνεται νομίζω πως πρέπει να αλλάξει. και αν δεν κάνω λάθος η εισηγήτρια τη ε, της έκθεσης στην Καθήλυνα Αρμόδια Επιτροπή έχει παρόμοια άποψη και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Τώρα, έχουν γίνει μεν κάποιες αλλαγές από τον εισηγητή του σχεδίου γνωμοδότησης, δεν ξέρω όμως αν είναι αρκετές. Εδώ βρίσκουμε πως ε, είναι προβληματικά τα σημεία για τις ε, επιγραμμικές πλατφόρμες, και σε γενικές γραμμές ε, να πω πως ε, δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι με αυτό το ε, σχέδιο γνωμοδότησης. Τα άρθρα 11 και 13 χρειάζονται επεξεργασία σημαντική. Ακριβώς διότι αυτή τη στιγμή συζητάμε μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτής της θητείας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πως ε, αυτό το θέμα αφορά όλους, πως έχουν εκφραστεί από όλα τα κρατημέλη τεράστιες ανησυχίες για το μέλλον των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και τεράστιες ανησυχίες για τη διατήρηση της ε, ακαιριότητας της νομοθεσίας. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω τα άρθρα 11 και 13 να επαναξεταστούν σημαντικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο και σε άλλους συναδέλφους. Ο κύριος Έλερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι απίστευτο. Δεν περίμενα ποτέ να δω την αριστερά να υπερασπίζεται ε, την καπιταλιστική Αμερική. Είναι κάτι που με εκπλήσει. Μετά από... Εντάξει, βέβαια έχουν περάσει και 20 χρόνια, 25 από την πτώση του τείχους, οπότε αλλάζουν πολλά πράγματα. Τώρα, Εδώ νομίζω πως ε, αναφέρθηκε πολύ σωστά ότι η εξόριξη δεδομένων πρέπει να περιέχει και μία εξαίρεση για την επιστημονική κοινότητα, για τους επιστήμονες οι οποίοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα ε, και επίσης ε, σε ό,τι αφορά τη χρήση για εμπορικού σκοπού, αναφέρθηκαν ορισμένε πολυεθνικέ, η Ford, α πούμε, η Google. Η Ford, να σα πω, πω ναι, μεν πουλά ε, προϊόντα, αλλά κάνει και τεράστια επιστημονική έρευνα από πίσω. Υπάρχει ένα τεράστιο επιστημονικό team το οποίο ε, εργάζεται πυρετοδός. Γι' αυτό δεν νομίζω πως ε, περιορίζοντας την πρόσβαση θα προστατευτούν τα δικαιώματα. Αντίθετα πιστεύω πως κινδυνεύει η πρόοδος της επιστήμης, της τεχνολογίας και πραγματικά μου φαίνεται απαράδεκτο να αναφέρετε την κοινωνία των πολιτών και να λέτε πως ε, οι μεγάλοι όμιλοι ασκούν πίεση, κάνουν λόμπι, να μιλάτε για την Google ως ε, τον ε, κακό. Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό. Τώρα, κάτι άλλο. Να υπενθυμίσω πως το Κοινοβούλιο ήδη έχει αποφασίσει μαζί με την Επιτροπή Πολιτισμού οι δημιουργικές βιομηχανίες, να το πω έτσι, η... που περιέχουν μικρούς επιχειρηματίες, δηλαδή μικρούς εκδότες, δημιουργούς, καλλιτέχνες. Ε, έχουμε συμφωνήσει να συζητήσουμε τη σημασία τους εδώ. Τώρα, πιστεύω πως με αυτήν την ε, πρόταση υπονομεύονται τα ε, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Υπονομεύονται οι ίδιοι οι μικροί δημιουργοί. Και πραγματικά, για να το πω ομά, νομίζω πως με αυτές τις προτάσεις πέφτει τσεκούρι σε ορισμένους ε, κλάδους, οι οποίοι εξαρτώνται άμεσα από ε, αυτό που συζητάμε και αφορούν μικρούς, μικρομεσαίους, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εμείς ε, φυσικά θέλουμε να υπερασπίσουμε την νόμιμη χρήση περιεχομένου από μικρούς ε, και ε, μικρομεσαίους δημιουργούς και να αποφύγουμε τη χρήση και τη συλλογή σκούπα, αν θέλετε, μαζικά συλλογή δεδομένων από μεγάλους ομίλους. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος Διακόπτη. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Έλερ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπλάνκο σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η πρόταση του εισηγητή ε, έχει βασικά στόχο την, ε, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά ε, και την εξόριξη στοιχείων. Εγώ θεωρώ πιο βάση με την πρόταση της Κομισιόν ε, παρόλα αυτά. Η πρόταση οδηγίας είναι ενδιαφέρουσα για, και σε πολλές στοιχείες τις οποίες δεν ανέφερε καν ο εισηγητής και που μας έχουν απασχολήσει επανελειμμένα σε αυτή την Επιτροπή. Πιστεύω δηλαδή συγκεκριμένα πως η οδηγία μας προσφέρει τη δυνατότητα να εξετάσουμε ένα θέμα κλειδί, όπως η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η, μετα... η... η... μεταβίβαση αξίας ε, όπως ας πούμε γίνεται στην νέα αγορά, την ψηφιακή, για τις ε, πνευματικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Πρόκειται για ένα ε, δικαίωμα το οποίο έχουν οι δημιουργοί για να μπορούν να αμευθούν για την εργασία τους, όπως ας πούμε το αναγνωρίζει η Ισπανική νομοθεσία. Ε, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας ε, και οι τροπολογίες τις οποίες εγώ θα υποβάλω θα ακολουθήσουν τη γραμμή που μόλις σας περιέγραψα. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ συνάδελφο, συνάδελφε. Η κυρία Γκάθα Γκέρμπα από την DG Connect εξ ονόματος της Κομισιόν. Thank uh, uh, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για την εργασία του για αυτήν την γνωμοδότηση και ευχαριστώ και όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Φυσικά θα επιμείνω στην εξόριξη στοιχείων και κειμένων γιατί αυτό ήταν το βασικό ζήτημα εδώ ε, και επίσης στις ανάγκες της επιστημονικής έρευνας. Είναι μια πολύ φιλόδοξη πρόταση που εμείς παρουσιάσαμε εδώ για την ε, εξόριξη στοιχείων και ε, κειμένων ξεπερνά τους ισχύοντες κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί πνευματικών δικαιωμάτων, copyright, αλλά και τις νομοθεσίες που ισχύουν στα περισσότερα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι σε αυτή μας την προσέγγιση περιλαμβάνουμε και ΣΔΙΤ, συνεργασίε, δηλαδή, εταιρικέ σχέσει μεταξύ ιδιωτικού και μη ιδιωτικού τομέα και δεν προβαίνουμε σε διάκριση μεταξύ εμπορικών και μη εμπορικών στόχων. Εμεί εστιάζουμε στην ανάγκη των ερευνητών και των ερευνητικών ιδρυμάτων, αλλά δεν προβαίνουμε σε διάκριση μεταξύ εμπορικών και μη σκοπών. Επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι δεν προσπαθούμε να επηρεάσουμε αγορές οι οποίες λειτουργούν σωστά ούτε τις άδειε που λειτουργούν σωστά. Γι' αυτό και έχουμε κάποιες ανησυχίες όσον αφορά την επέκταση του πεδίου εφαρμογή ε, που προτείνει ο εισηγητής, που πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε στην ε, ορθή και ομαλή λειτουργία των αγορών. Θέλουμε λοιπόν να εκφράσουμε αυτή μας την ανησυχία σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Κύριε καθηγητά, ακούστηκαν διαφορετικές απόψεις ε, και εντός της Επιτροπής Ήτρε. Θα χρειαστεί λοιπόν να αγωνιστούμε πώς θα βλέπετε τα πράγματα Κοιτάξτε, η συζήτηση μόλις επιβεβαίωσε την άποψή μου ότι σε αυτό το θέμα υπάρχουν τόσο πολλά συμφέροντα και τόσο πολλά ε, επιχειρήματα που ακόμα και εντός της ίδιας μας της Επιτροπής δεν συμφωνούμε απόλυτα. Ανέφερα ότι το άρθρο 11 είναι επίμαχο και το 13 επίσης και δεν αναφέρθηκα καν στα θέματα γιατί αυτό, ε, των άρθρων αυτών, γιατί αυτά ξεπερνούν τις δικές μας αρμοδιότητες, αλλά θέλω να υπερασπιστώ τη θέση μου. Συνάδελφοι, εγώ μίλησα για την κατάσταση, ανέφερα αυτά που είχα υπόψη μου και όντως ο καθένας έχει τη δική του προοπτική. Εγώ έχω την προοπτική ενός ε, ε, επιστήμονα. Και τα πράγματα έχουν ως εξή. Αν έχει κανείς νόμιμη πρόσβαση στο περιεχόμενο, σημαίνει ότι το την πληρώνει, αλλά δεν μπορεί να δει το περιεχόμενο αυτό με ηλεκτρονικό τρόπο. Και αυτή η κατάσταση είναι τελείως παράλογη. Κάποιος αγοράζει λοιπόν το περιεχόμενο και είτε είναι επιστήμονας είτε είναι οτιδήποτε γιατί στη Γερμανία έχουμε αυτό το private gelaten, αυτού τους, τους ιδιώτες ε, επιστήμονες που έχουν δημιουργήσει και έχουν συμβάλει πολύ στην επιστήμη. Γιατί λοιπόν οι άνθρωποι εκτός των επιστημονικών Ινστιτούτων να μην μπορούν να κάνουν εξόριξη στοιχείων, γιατί να πρέπει να πληρώσουν για επιπλέον λογισμικό, δεν μπορώ αυτό να το καταλάβω. Το ίδιο με τη διάκριση μεταξύ εμπορική και μη χρήση. Είναι σχεδόν αδύνατο να το ερευνήσουμε αυτό, γιατί το μεγαλύτερο τμήμα τη επιστημονική έρευνα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εμπορικά στη βιομηχανία αργότερα. Έχουμε ένα ολόκληρο τομέα της βιομηχανίας που καταλαβαίνω θέλετε να τον υπερασπιστείτε, που Έχουμε και τους εκδότες των επιστημονικών περιοδικών ή βιβλίων των οποίων συχνά το επιχειρηματικό μοντέλο βασίζεται σε δημόσια κονδύλια, γιατί περισσότεροι ε, επιστήμονες στην Ευρώπη χρησιμοποιούν δημόσια χρηματοδότηση και συχνά χρησιμοποιούν ε, το τα πραγματικά τους δικαιώματα για να περιορίσουν την πρόσβαση ε, στο περιεχόμενό τους, πράγμα το οποίο είναι σημαντικό και χρήσιμο για να βοηθηθούν οι επιστήμονες να δημιουργήσουν πολιτιστικό ε, περιεχόμενο. Ευχαριστώ. Είμαι εδώ λοιπόν και είμαι έτοιμος να ε, αγωνιστώ. 28 Μαρτίου 2017 είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών στις 12. Θα ψηφίσουμε το Μάιο στην Ήτρα και θα είμαστε στην ώρα μας γιατί ε, είναι μια γνωμοδότηση που απευθύνεται στην Επιτροπή Γιούρη. Και η ψηφοφορία εκεί θα γίνει από όσο γνωρίζω τον Ιούλιο. Να περάσουμε λοιπόν στις ψηφοφορίες. If you could uh, take a seat, dear colleagues, ladies and gentlemen. Καθίστε παρακαλώ, κυρίες και κύριοι. Uh, uh, well, moment. Uh, dear colleagues, ladies. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, ε, κυρίες και κύριοι, έχω ένα λεπτό καθήκον, μια λεπτή ανακοίνωση για όλους μας. Καθίστε παρακαλώ πολύ. I've uh, Έχουμε ε, μια, όπως σας είπα, θλιβερή ανακοίνωση. Ακριβώς πριν από ένα χρόνο ήμασταν όλοι μας μάρτυρες, ε, όλοι μας όσοι ζούμε και εργαζόμαστε στις βρυξελλες τεσσερις τέσσερις-πέντε μέρες την εβδομάδα, Ζούμε εδώ στην πόλη μα. είναι η πόλη μα οι Βρυξέλλε και ήμασταν μάρτυρες μια φρικτής τρομοκρατική επιθέση ακριβώς πριν από ένα χρόνο το πρωί. Όλοι θυμόμαστε πάρα πολύ καλά εκείνη την ημέρα. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να ε, θυμίσουμε τα θύματα της ε, τρομοκρατικής επίθεσης του 2016 στις Βρυξέλλες και για να δείξουμε την αλληλεγγύη μας με τις οικογένειες ε, αλλά και μεταξύ μας. Τις οικογένειες των θυμάτων αλλά και μεταξύ μας ε, που είμαστε εδώ στις Βρυξέλλες, δραστήριοι και πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος για να δείξουμε ότι το στιμόμαστε και να δείξουμε την αλληλεγγύη μας είναι να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή.

put your cards into the slot. Παρακαλώ, τοποθετήστε τις κάρτες σας στις οπές και θα κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία όσοι ήθιστε. Άρχεται. Παρακαλώ, χρησιμοποιήστε ένα από τα κουμπιά. Uh, has anybody όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Νομίζω ότι όλα τα μηχανήματα λειτουργούν, οπότε ας προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Έχουμε κατάλογο ψηφοφορίας ε, για το σχέδιο έκθεσης για την πρόταση απόφασης ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συμμετοχή της Ένωσης στην εταιρική σχέση στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου, που αποκαλείται πρίμα. Η Σοφία Σακοράφα της Γκουε ήταν η συγγήτριά μας. Λοιπόν, συμβιβαστική 1, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται NV15 υπέρ κατά αποχές έλεγχος NV15 I close the vote. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 115 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. ΕΝΒ 18 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. ΕΝΒ 21 υπέρ κατά αποχές εκρίνεται ε, 126 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές γκρίνεται 23 είναι unblock τώρα 23, 24, 26, 27 28, 29, 30 41, 42, 43. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 25 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Α, ψηφοφορία τώρα unblock είναι η 129, 197 και η NV22. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. NV23 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται νομίζουμε. Ας ελεγξουμε Εν NV23. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εν 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 130 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ. no. Okay. Sorry. Block. Πρόεδρο, συγγνώμη. Έχουμε πρώτο μπλοκ της Envy. Είναι δύο τροπολογίες, 25 και 26. Αν μπλοκ υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτονται. 31 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, η 32 υπέρ. Α, θέλετε έλεγχο. Έλεγχο για την 31. 31 ηλεκτρονικός έλεγχος. Και πέρας πληροφορία, εγκρίνεται. 32 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NV28 υπέρ κατά για να δούμε έλεγχος NV28 τέλος της ε, ψηφοφορίας ε, απορρίπτεται 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV36 υπέρ. NV36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μάλιστα. Θέλετε να το ελέγξουμε, να το ελέγξουμε. MV36. I close the vote. Rejected. Rejected. Απορρίπτεται. 162. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ναι, να το ελέγξουμε. 162. 162. 162 ελέγχουμε. Ηλεκτρονικά τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται. NV40 υπέρ. Κατά. Ε, έλεγχος ηλεκτρονικός. NV40. I close the vote. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 167. Αποκινούμε την προφορική τροπολογία. Και υπάρχει γενική συμφωνία για την ε, προφορική τροπολογία από ό,τι ξέρω. Α ψηφίσουμε λοιπόν την 167. Μαζί με την προφορική. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 185 και 186 από κοινού. Υπέρ, κατά, αποχές, ΕΝΒΙ NV44, υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 188, unblock, 44, 45, 188, 189. Βλέπετε τώρα τις τροπολογίες. Είναι πολλές. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μπλοκ 3. 192 και το καθεξής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Όλα από κοινού. 192, 200. Και η ένβη 13. Όχι. Καταπίπτει. Είναι μόνο 192 και 200. Δύο λοιπόν τροπολογίες από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ένβη 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 145. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 5, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 53, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 6, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. NV1, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 56. Πέρας. Εγκρίνεται η 56. Παρακαλώ, επί της διαδικασίας η NV45 ήταν αυτή. Νομίζω ότι δεν είδαμε την ε, NV45. NV45 λέτε. Για να τη βρω μια στιγμή. Η ένδυ 45 είναι στη σελίδα 17. Σωστά. Καταπίπτει. Επειδή εγκρίθηκε το Block Vote 2. Η σελίδα 16 θα το βρείτε αυτό. Εκεί λοιπόν αναγράφεται ότι η NV45 καταπίπτει εάν εγκριθεί ε, η ψηφοφορία κατά τμήματα στο σημείο 2. Εντάξει, είμαστε τώρα στην 56. Α, εγκρίθηκε. Τροπολογία 58, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 59, υπέρ. Να ελέγξουμε την 58. Από την αρχή. 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ξεκάθαρα απορρίπτεται. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. NV3. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές Ας ελέγξουμε. Την 60. Πέρας. Απορρίπτεται. Τρία. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Δεν είναι ξεκάθαρο. Πέρας. Απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. NV7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εντάξει, να ελέγξουμε. Την ένβη 7. Πέρασε. Εγκρίνεται. Α, σας ευχαριστώ που το επισημάνατε. Ένβη 8, υπέρ. Κατά. Αποχές, ας ελέγξουμε και πάλι. Πέρας. Εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 73 και NV9 από κοινού υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά αποχές. Ας ελέγξουμε την 75. Πέρας. Απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Την 79. Πέρας. Απορρίπτεται. 80. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε και πάλι. Την 80. Πέρας. Απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές ας ελέγξουμε την 87. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα, 83 και 84. Α, 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 89 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε την 89. Πέρας. Απορρίπτεται αυτή τη φορά. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 90. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε. Την 9 πέρας ψηφοφορίας. Α, συγγνώμη, δεν ήταν ξεκάθαρο. Εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα δύο τροπολογίε από κενού, 95 και 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 105 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13 καταπίπτει. Citations. 47 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Τη 47 πέρας. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Είμαστε όλοι εδώ, λέει ο Πρόεδρος. Και πάλι όμως έχουμε ένα παραπάνω από το ΕΛΚ. Τι να κάνουμε τώρα. Α, εντάξει τώρα. Ευχαριστώ. Είδες ή ήξερες τι να κάνεις. Γιατί μία ψήφος είναι σημαντική. Εγκρίνεται λοιπόν 48 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 49 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση για το σχέδιο έκθεσης. Με ονομαστική κλίση παρακαλώ. Πέρας. «55 υπέρ, 7 κατά, Και τώρα για τις διοργανικές διαπραγματεύσεις και πάλι με ονομαστική κλίση παρακαλώ ψηφίζουμε. Πέρας. 59 ψήφοι υπέρ, μία κατά. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία εισηγήτρια, όλους τους κοιόδης, όλους εσάς συνάδελφοι. Ας περάσουμε τώρα στην δεύτερη ψηφοφορία, σχέδιο γνωμοδότησης. Δεσμευτικές αιτήσει μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα κάτω μελη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική ενεργειακή ένωση. Ο συνάδελφος Μπένετιτ Γιάβορ είναι εισηγητής. Ας περάσουμε στις ψηφοφορίες. Συμβιβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 79. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 80. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 82. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 82. Πέρας. Απορρίπτεται. 83. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε την 83 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Να αρχίσουμε από την αρχή, καλύτερα. Εφόσον το θέλετε. Άρχεται η ψηφοφορία. Από την αρχή. Την 83, τροπολογία 83. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. να ελέγξουμε τη συμβιβαστική 2. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 96-154 και 159. Τρεις λοιπόν μαζί, υπέρ. Κατά. Καλύτερα να ελέγξουμε ηλεκτρονικά τις τρεις αυτές τροπολογίες μαζί. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνονται. Περνάμε στη συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Επαναλαμβάνω. Η 97... Α, συγχωρείτε συνάδελφοι, με συγχωρείτε. Πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 97. Αφού ψηφίσουμε τρεις ε, τροπολογίες μαζί. Περνάμε στην 97, όχι στη συμβιβαστική. 97 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την συμβιβαστική 3. Πέρας. Εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θα την ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 122. Πέρας. Απορρίπτεται. 107. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 106. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 105. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 109. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 110. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 108. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 111. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε την 111 ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά τη Συμβιβαστική 4. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεκαοχτώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 140. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 141. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 142. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 145. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 146 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 147 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 148 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 21, 149, 150 και 171. Τέσσερι τροπολογίες μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 151 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 158 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 24. Πέρας. Εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε την 25. Πέρας. Απορρίπτεται. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 167. Πέρας. Απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. 26. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Την 27. Πέρας. Εγκρίνεται. 28. Υπέρ. Κατά.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 Ελέγχουμε. Τη 40. Πέρας. Απορρίπτεται. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Α... Ας ελέγξουμε. Ας ελέγξουμε. Τη συμβιβαστική 11 πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Την 6 Πέρας ψηφοφορίας. Θέλετε ξανά. Μάλιστα. Τροπολογία 6. Καταλαβαίνω πως χρειάζεστε και άλλο χρόνο. Πάμε από την αρχή λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Αρχίζουμε από την αρχή. Τροπολογία 6. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Με ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα από πριν. 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Ευχαριστώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Δεν ήταν σαφές. Ελέγχουμε την 67. Ναι, η 66 καταπίπτει. Τώρα ψηφίζουμε την 67. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Δεν ψηφίζεται, συνάδελφοι. Δεν βλέπω τίποτα εδώ. Δεν βλέπω χέρια. Δεν ψηφίζεται. Τροπολογία 68 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Λυπάμαι που σας το κάνω αυτό. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση για το σύνολο σχεδίου έκθεσης. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 35 ψήφοι υπέρ, 28 κατά. Εγκρίνεται η έκθεση. Περνάμε στην επόμενη έκθεση. Ευρωπαϊκά πρότυπα και εφαρμογή του κανονισμού 1025, κάθετος 2012. Εισηγητής ο Χάνς Όλαφ Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά. Αποχές ελέγχουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές Α ελέγξουμε και ψηφίστε παρακαλώ συνάδελφοι τη την τροπολογία 9. Πέρας. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 11. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Για να είμαστε σίγουροι. Πέρας. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε τη 12 ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά τη 14. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε την 55. Πέρας. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε την 57. 57. Πέρας. Απορρίπτεται. 60. Όχι. 59. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε την 109. Πέρας. εκρήματα. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε την 72. Πέρας. Απορρίπτεται. 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 75. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η προστίκη στη συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές ας ελέγξουμε. Συμπληρωματική πρόσθετη στην συμβαστική 8. Πέρας. Απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 102 υπέρ. Με συγχωρείτε, λέει Τροπολογία 100. Υπέρ κατά αποχές. Ας την ελέγξουμε. 100. Πέρας. Απορρίπτεται. 101. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 102. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προσθήκη στη συμβαστική 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ, κατά αποχές Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 107. Πέρας. Απορρίπτεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. 115. Πέρας. Εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 118 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε την 118. Πέρας. Απορρίπτεται. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ. Κατά. Α... Εγκρίνεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 129 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε την 129. Πέρας. Απορρίπτεται. 130. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ενομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Όπου, Χάνσόλαφ Χένκελ, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε εσά, συγχαρητήρια σε όλους τους κοιόδους συζητητές και περνάμε στην τελευταία ψηφοφορία για σήμερα. Σχέδιο γνωμοδότησης για την συνεργατική οικονομία. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκίνεται. 49 ε, υπέρ κατά αποχές εγκίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκίνεται. Συμβαστική 10 α υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10B υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 87, όχι, 87. 90 87 τμήμα 2. Είναι στη σελίδα 9. 87 τμήμα 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε. Ελέγχουμε. 90. Και τέλος της ε, ψηφοφορίας. Ε, εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ κατά αποχές 111 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική. Όχι αυτή την έκθεση μόνο, αλλά και για δύο μέρες. για τη σημερινή μάλλον ψηφοφορία. 53 υπέρ. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια στον συγκεκριτή. Ευχαριστώ όλους. Four reports. Okay, let us go to the next Ας περάσουμε στα επόμενα σημεία. For, for, for... Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλουμε να ξεκινήσουμε σε δύο-τρία λεπτά. Παρακαλώ, όσοι να καθίσετε, καθίστε. Και να μην, ε, και να μην συζητάτε πια φωναχτά. Α, παρακαλώ, εγώ προτιμώ να μείνετε, βεβαίως, εντός της αίθουσας. Okay. Hello. No, we start immediately. Ναι, όχι, ξεκινάμε αμέσω. Πέντε λεφτά, όχι ούτε πέντε λεφτά. Any, any Uh, uh, dear colleagues, uh, member of our Αγαπητοί συνάδελφοι, ζήτησα ένα παλαιό μέρος ε, της Επιτροπής μας να προεδρεύσει, γιατί τώρα πρέπει να πάω κάπου αλλού. Είμαι ευγνώμων λοιπόν στον Πολ Ρούμπικ, που είναι παλαιό και σπουδαίο μέλος της Επιτροπής να συνεχίσει ε, εκείνος την Προεδρία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο. Για τα καλά του λόγια, ναι, εννοεί ότι είμαι παλιός στην Επιτροπή, όχι ότι είμαι ο κυριότερος. Και είναι πολύ λοιπόν σημαντικό να ε, Κάνουμε αυτήν την συζήτηση για τον Ευρωπαϊκό Κώδικα, Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα στα πλαίσια της ψηφιακή αγοράς και γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι πάρα πολύ που η κυρία Πιλάρ Ντακαστήγιο είναι εισηγήτρια, διότι ασχολείται πολλά χρόνια με, την, ε, με το ψηφιακό θεματολόγιο. Έχουμε 40 λεπτά στη διάθεσή μας για αυτό το θέμα και θα αρχίσω δίνοντας το λόγο στην Πιλάντε Καστίγιο ως εισηγήτρια του ΕΛΚ. Έχετε πέντε λεπτά χρόνο για να παρουσιάσετε το θέμα αυτό. Παρακαλώ, Πιλάρ. Thank ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να αρχίσω τονίζοντας ότι από την αναθεώρηση του 2009 η αγορά έχει αλλάξει δραματικά. Έχουν εμφανιστεί και άλλοι παράγοντες και γενικά οι υπηρεσίες έχουν αυξημένη σημασία. Η συνδεσιμότητα και τα μήκη κύματος σημαίνουν υψηλή ανάγκη για περισσότερη τεχνολογία. Ε, ο ιδιωτικός τομέας θα κληθεί να καλύψει την πλειοψηφία του ε, ποσοστού αυτού. Έτσι θα εξασφαλιστεί η προβλεψιμότητα και η ανάληψη του κινδύνου για μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Η πρόταση της Κομισιόν να προσθεθεί υποδομή στην πυρήνα του πλαισίου, κατά τη γνώμη μου, είναι η σωστή προσέγγιση. Επενδύσεις, ανταγωνισμός, κανονισμοί θα πρέπει να αποτελέσουν έναν ε, ενάρετο κύκλο για την ανάπτυξη ε, δικτύων υψηλής ε, ε, χωρητικότητας για τους αρμόδιους για τις προσλήψεις. Τώρα όσον αφορά την πρόσβαση, πιστεύω πως η προσέγγιση του ανταγωνισμού που βασίζεται στη σημαντική ισχύ της αγοράς θα πρέπει να παραμένει στην καρδιά της προσπάθειας. Το πλήρες, η πλήρης εργαλειοθήκη θα πρέπει επίσης να επιτρέπει και να παραμένει ε, στα χέρια των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Ωστόσο, στηρίζω την πρόταση της Κομισιόν, μέσω της οποίας οι, τρέχο, ισχύοντες στόχοι θα καλυφθούν από τους νέους στόχους συνδεσιμότητας. Σε αυτό το πλαίσιο έχω υποβάλει προτάσεις ε, όπως ε, ε, η αναθεώρηση ας πούμε της, ε, η διαδικασία ε, αναθεώρησης αγοράς για πολύ δυναμικές αγορές η παράταση στα 5 χρόνια, η επέκταση μάλλον στα πέντε χρόνια θα μπορούσε να καταλήξει σε έναν κανονισμό ο οποίος επιμένει πέρα από τα όσα είναι απαραίτητα και Εάν ε, στις συγκεκριμένες αγορές ε, γίνει νέα ανάλυση αγοράς, όπως ε, θα πρέπει να γίνεται κάθε τρία χρόνια όπως ισχύει σήμερα. Τώρα, γεωγραφική υπηρεσία. Νομίζω πως η επιβολή υποχρέωσης στους operators για να παρουσιάσουν συγκεκριμένη πρόβλεψη με πιθανή επιβολή κυρώσεων είναι δυσανάλογο κατά τη γνώμη μου και δεν λαμβάνει υπόψη αρκούντος τις αποφάσεις που λαμβάνονται με ε, ε, τον ολισμό στην αγορά. Τώρα, για τις διευκολύνσεις θα πρέπει να διευκολύνουμε την ε, ανάπτυξη εναλλακτικών δικτύων στις ε, αεροκατοικημένες περιοχές. Ωστόσο, αυτή η υποχρέωση δεν θα πρέπει να ισχύει εάν ε, εάν υπάρχει πρόσβαση και σε άλλα δίκτυα. Και όλα αυτά θα πρέπει να υπόκειται στην δυνατότητα σύναψη συμφωνιών για πρόσβαση με πάντοτε ένα άνοιγμα προς την, ε, τον ανταγωνισμό. Τώρα, το φάσμα. Το φάσμα είναι σημαντικός πόρος. Α, προς, αυτό, εγώ στηρίζω την θέση τη διαρκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Ε, Επίση υπεστηράζομαι την ε, μίνιμουμ διάρκεια της άδεια για 30 χρόνια για τα προηγμένα ε, δίκτυα. Η αυξημένη διάρκεια συνοδεύεται από πιο αυστηρές απαιτήσει που στόχο έχουν τη χρήση, την αποτελεσματική χρήση του και την ε, αποδοτική χρήση του ε, φάσματος με μηχανισμούς ε, χρησιμοποίησε το ή, να, ή χάσε το για τη βέλτιστη χρήση, για τις, τη βεβαιότητα των επενδύσεων. Έχω προτείνει τροπολογίε να εξασφαλίσουμε ότι οι προτάσεις για τα ατομικά δικαιώματα δεν θα αλλάζουν χωρίς συμφωνίες. Επίσης, υποχρέωση παροχής υπηρεσίας, ενίσχυση της εμπορίας και να εξασφαλίσουμε ότι μια δίκαιη τιμή θα βασίζεται στη σωστή αξιολόγηση των συνθήκων της αγοράς. Και τέλος, για να έχουμε συγκεκριμένους πόρους για τη βελτίωση και τον συντονισμό, του συντονισμού ανάμεσα στα κάτι μέλη, προτείνω να ενισχυθεί ο ρόλος της ομάδας πολιτικής για το φάσμα. Έχουμε δίκτυα με πολύ ψηλές δυνατότητες και πιστότητα. Αναγνωρίζω ότι το 5G είναι η τεχνολογία του μέλλοντος. Αναγνωρίζω και ότι η τεχνολογική ουδετερότητα του δικτύου πρέπει να είναι ε, η βασική μας αρχή, δικτύου υψηλής ε, ταχύτητας. Και γι' αυτό προτείνω και ένα δυναμικό ορισμό που βασίζεται στη δυνατότητα των δικτύων να ανταποκριθούν στι ανάγκες για, για συγκεκριμένη μάλλον χρήση και να συνδέονται όλα αυτά και με παραμέτρους απόδοσης ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι συνδεσιμότητας μέχρι το 2025. Ε, προτείνω να συμπεριληφθούν όλες οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας με ένα συγκεκριμένο κατόφλι για τις μικρές ε, δυνατότητες. Αυτή είναι η σύντομη σύνοψη του σχεδίου εκθεσής μου και τώρα ε, προσβλέπω στις δικές σας ε, παρατηρήσεις και απόψεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Uh, next one is minutes uh, for every Δύο λεπτά για κάθε σκιώδη. Πρώτα έχουμε το Σοσιαλιστές Κομπούλα Νάτρι uh, πρέπει να πω ότι είναι πολύ επαγγελματική αυτή η εργασία και σηματοδοτεί το τέλος των 146 τροπολογιών. Βέβαια δεν μπορώ να... Δεν θα σχολιάσω κάθε μία τροπολογία χωριστά, αλλά ε, εδώ έχουμε υποσχέσεις ε, για την οικονομία μας και τώρα κοιτάμε το πλαίσιο. Το πλαίσιο δεν θα πρέπει να μας φοβήσει για την επίτευξη αυτού του στόχου. Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι βέβαια και οι σωστέ επενδύσεις, γιατί χωρίς δρόμους δεν έχουμε και ε, σωστές, σωστές ε, μάλλον, δεν μπορούν να κυλήσουν και τα ποδήλατα ή τα αυτοκίνητα. Ε, Πιστεύω πως ο ανταγωνισμός ε, ε, οδηγεί, καθοδηγεί τις επενδύσεις ε, και όλο ένα και περισσότερο έχουμε σήμερα και, και άλλες καινοτομίες και αυτό παίζει ρόλο σε κάποιους τομείς όπως αυτός εδώ. Σημαντικός είναι ο ρόλος και των τελικών χρηστών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και της βιομηχανίας, εάν θέλουμε να αλλάξουμε προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πρέπει να αλλάξουμε και πορεία. Και ερώτησή μου προς την εισηγήτρια είναι Ποιος είναι ο νέος ορισμός για τα δίκτυα πολύ υψηλής ε, χωρητικότητας και ταχύτητας. Εγώ ε, πιστεύω πως δεν θα πρέπει να στηριχτεί η βιομηχανία για κάτι το παλιό. Αναφέρθηκε το IDSL. Αυτό είναι ήδη ξεπερασμένο. Ξέρουμε πως οι χώρες έχουν διαφορετικές ε, ε, συνθήκε, αλλά αφού είναι πίσω δεν χρειάζεται να τι χρηματοδοτήσουμε για αυτή την τεχνολογία. Αν έχει κάνει βουνά είναι, ε, είναι πιο δύσκολο από ότι αν έχει μικρή πυκνότητα. Αλλά μετά είδαμε και νεοφερμένους όπως οι Λετονοί, οι Λιθουανοί, οι Ρουμάνοι. Ε, δεν, έχει να κάνει με το αν είσαι πλούσιος ή και για το φάσμα η συγκήτρια είπε πω χρειάζεται για τις νέε τεχνολογίε αλλά υπάρχουν και τροπολογίες που αφαιρούν την υποχρέωση για μοιρασιά. Γι' αυτό και θέλω να δούμε πώς στο μέλλον θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις μελλοντικέ επενδύσεις. Ευχαριστώ και εγώ. Ε, ECR. Να σας συγχαρώ για την επανεκλογή σας ως Αντιπρόεδρο στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ και για την προσωπική σας ε, στήριξη. Είμαι... Αισθάνομαι μεγάλη τιμή που μπορώ να προσφέρω βοήθεια σε αυτήν τη σημαντική επιτροπή, την ΣΤΟΑ. Εκτιμώ την εργασία της Πλάρτε Καστήλου. ήταν πολύ επαγγελματική και η έκθεσή της είναι πολύ εμπεριστατωμένη παρότι πολυτεχνική. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα περίπλοκο πλαίσιο να φτιάξουμε, μάλλον να, να προσφέρουμε την ε, νομική σταθερότητα και βεβαιότητα και να αναλύσουμε μεμονωμένα τα μέτρα που προτείνει η Κομισιόν. Εκείνη έχει μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη σε αυτό το τομέα και αυτό το εκτιμώ πάρα πολύ. Φυσικά έχω κάποια σχόλια. Θα προτιμούσαμε ίσως κάποιες συγκεκριμένες λύσεις και θα ήθελα αυτές να τις αναφέρω. Αυτή την έννοια της ε, υψηλής χωρητικότητας πρέπει να βρούμε έναν συγκεκριμένο αλλά ρεαλιστικό τρόπο να προχωρήσουμε και είναι προτείνει λύσεις ε, που οδηγούν προς μεγαλύτερη τεχνολογική οδητηρότητα που είναι σημαντική όμως αμφιβάλλω κάπως για τον ορισμό της απεριόριστης χρήσης γιατί θα χρειαστεί αυτό να το συζητήσουμε. Είναι επίσης μια ενδιαφέρουσα λύση για την ανάλυση της αγοράς. Εγώ είμαι υπέρ της τη της περίοδου ανάλυσης αγοράς στα πέντε χρόνια αλλά και το, η πρόταση της εισηγήτριας είναι λογική. Τώρα, για τα επενδυτικά πρότυπα ε, νομίζω πως θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να βρούμε σωστή ισορροπία και να επενδύσουμε σε μια ουδέτερη ε, στάση. Να μην σταθούμε εμπόδιο δηλαδή στις επενδύσεις ε, Επίσης, ε, ενδιαφέρουσες είναι άλλες ε, διατάξεις, ότι δηλαδή βασικά θα πρέπει να παραμείνει η Επιτροπή δεν θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί στην εναρμόνιση αυτού του τομέα. Όσον αφορά την επέκταση της αδειοδότησης στα 25 χρόνια, είναι πολύ μακρά περίοδος αυτή. Είμαι υπέρ πιο ευέλικτων λύσεων. Προσβλέπω λοιπόν στην συζήτηση αυτής της συζήτησης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. επόμενη είναι η κυρία Κάλλας από την Άλντε. Ευχαριστώ πολύ και για την έκθεση. Είναι πολύ σημαντική, γι' αυτό επειδή είναι και εκτενές κείμενο, δεν θέλω να επιστρέψω λεπτομέρειε, λεπτομέρειες. Πρώτα απ' όλα, προτεραιότητα της ομάδας μου με αυτή την αναθεώρηση του πλαισίου ε, είναι η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς η ρυθμιστική σύγκληση δεν αρκεί αν θέλουμε μια αγορά που θα μας φέρει αγορές κλίμακας και θα ενισχύει τον ανταγωνισμό για να προσελκύει και τις επενδύσεις στα δίκτυα που είναι ο γενικός μας στόχος. Παρότι για τα καθορισμένα ε, δίκτυα η κατάσταση είναι πιο πολύ εθνική, ακόμα και τοπική. Γι' αυτό Χρειαζόμαστε ένα περιθώριο ευελιξία και για το φάσμα και για τι υπηρεσίε που είναι πολύ πιο διασυνοριακέ στη φύση του. Η έλλειψη τη ενιαία αγορά είναι περισσότερο ζήτημα πολιτική βούληση και όχι τεχνολογία ή γεωγραφία. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Τώρα για τους βασικούς ε, στόχους ε, του κώδικα που αναφέρει η Επιτροπή, όντω ε, τα δίκτυα πολύ ψηλή ικανότητα είναι ένα στόχο, δεν ξέρουμε πώ μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ε, ε, τον ανταγωνισμό. Πρέπει λοιπόν να διαφυλαχθεί ο ανταγωνισμός, αρκεί να υπάρχουν φορείς που ε, δραστηριοποιούνται και στη χονδρική και στη λιανική. Αν πάμε στο, στην αποσύζευξη χονδρικής και λιανική τότε θα ήταν πολύ χαμηλότερη ε, η ανάγκη ρύθμιση. Όμω δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Στη νέα προσέγγιση προτείνει η εισηγήτρια για να διαχωρίσουμε τι υπόλοιπε διατάξει για τα δίκτυα πολύ ψηλή ικανότητα. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει ακριβώ ποιε θα είναι οι προεκτάσει για τα υπόλοιπα δίκτυα. Εφόσον ε, πρόκειται για θεμελιώδη στόχο, ε, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να ισχύει για πολλά τμήματα του κώδικα, οπότε διαρωτώ με γιατί να μπει σε αυτό το συγκεκριμένο τμήμα. Ε, υπάρχει πόνοια από τον τίτλο αυτό ότι ο μοναδικό τρόπο να επενδύσουμε στα δίκτυα πολύ ψηλή ικανότητα ε, είναι μέσω τη ε, συνεπένδυση, co-investment, και εγώ διαφωνώ. Για το φάσμα ε, θέλει να παρατείνει τη διάρκεια στα 30 έτη. Δεν συμφωνώ με αυτή την παράταση γιατί ουσιαστικά μπορούν να υπάρξουν και νέες τεχνολογικές καινοτομίες και επιλογές για, για την καλύτερη χρήση του φάσματος. Πρέπει να συνδέεται και με ισχυρέ διατάξεις σε δευτερογενούς αγοράς και πάλι για τη χρήση του φάσματος για να αποφύγουμε τέτοιου είδους ε, ε, παγίδες. Για τους ορισμούς τώρα το μεγαλύτερο τμήμα των αρμοδιοτήτων ε, υπάγεται στην ΙΜΚΟ. Υπάρχουν ακόμα όμως ε, ζητήματα που εμπίπτουν ε, στον τομέα αρμοδιοτήτων της ΣΥΤΡΕ. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει κάποια διευκρίνηση για να συνάδουμε και με τις άλλες συναφείς οδηγίες. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σολεμόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ συμφωνώ προφανώ ότι είναι πολύ σημαντικό το έγγραφο και ότι η συγγήτρια ε, εκπώνησε ένα πολύ καλό προσχέδιο. Νομίζω ότι πολλέ ε, τροπολογίε ξεκαθαρίζουν, αποσαφηνίζουν το κείμενο ε, σε σχέση με το αρχικό κείμενο της Επιτροπής, οπότε είναι σωστή αυτή η κατεύθυνση. Έχω ορισμένε παρατηρήσει να κάνω τώρα. Πρώτον, οι ορισμοί που μα δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι είναι μια υπηρεσία τηλεπικοινωνία. Είναι παροχημένοι αυτοί οι ορισμοί, πρέπει να τους επικαιροποιήσουμε και να τους προσαρμόσουμε στη σημερινή κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια κοινή ε, αντίληψη για το τι θέλουμε να ρυθμίσουμε ακριβώς. Αλλιώς μπορεί να επηρεάσουμε και πράγματα που δεν θέλουμε να αγγίξουμε. Δεύτερον, για τις υποδομές και τις υπηρεσίες. Νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε από πλευρά συνταγωνισμού στις υποδομές και όχι τόσο στη λιανική. Πρέπει να δώσουμε έμφαση σε αυτό και όχι αυτό που σημαίνει αυτή τη στιγμή στην έκθεση και αυτό με φέρνει στο τρίτο σημείο, τα δικαιώματα χρήσης. Υπάρχει κάθετη ολοκλήρωση σε όλο τον κλάδο. Πρέπει τώρα λοιπόν να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των χρηστών, τι συμβαίνει με τα ε, δεδομένα του καθενός, ε, τι επιτρέπουμε να συμβεί με τα προσωπικά δεδομένα, ε, όροι και προποθέσεις, τέτοιου πράγματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν να ασχοληθούμε πιο συγκεκριμένα με αυτά τα ζητήματα. Και κάτι τελευταίο για το φάσμα, ούτε εγώ Είμαι πεπισμένο ότι η παράταση της διάρκειας θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό ε, και θα δώσει ωφέλη για τους ε, τελικούς χρήστες. Αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι δεν ε, είμαστε πεπισμένοι για την χρησιμότητα της παράτασης των αδειών. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα να το λόγο η επόμενη. Ε, συνάδελφοι, για ένα λεπτό ο καθένας. Ε, αρχίζουμε με τον κύριο Μπλανκολόπες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια και για την ταχύτητα με την οποία εργάστηκε. Ε, συμμεριζόμαστε τις ε, αρχές της και θεωρούμε και εμείς ότι τα δίκτυα πολύ υψηλής ικανότητας, υψηλής ικανότητας είναι σημαντικός στόχος μαζί και με την ενίσχυση τη εσωτερική αγορά και ούτω καθεξή. Ό,τι αφορά την προστασία του καταναλωτή, δεν συμφωνώ με την πρόταση τη Κομισιόν να έχουμε μια μέγιστη εναρμόνιση, γιατί αυτό σε κάποιε περιπτώσει μπορεί να σημαίνει και την ε, απομείωση ε, του επίπεδου προστασία, ιδίω σε ό,τι αφορά τι καθολικέ υπηρεσίε ε, να μην περιοριστούμε μόνο στην κρατική χρηματοδότηση, να γίνει και μέσω ιδιωτικών επιχειρήσεων. Η συγγετρία προτείνει τη διαμόρφωση ενό ειδικού τμήματο για τα δίκτυα ε, πολύ υψηλή ικανότητα. Εγώ δεν είμαι βέβαιο. δεν λέω ότι είμαι και αντίθετο, αλλά έχω κάποιες επιφυλάξει. που προκύπτουν από κάποιες από τις διατάξεις, αλλά και κάποιες από τις παραλήψεις σε ό,τι αφορά όλες τις ηλεκτρονικές τηλεπικοινωνίες, ψηφιακές ή όχι. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο χρειάζεται σε βάθος ανάλυση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρόιλ έχει το λόγο. Είναι σχεδόν αδύνατο να μιλήσει κανείς μόνο ένα λεπτό για κάτι τέτοιο. Ε, όταν μιλάμε για ένα τόσο σημαντικό θέμα, λοιπόν, πρέπει καταρχάς να μιλήσουμε για ε, το πώς θα δώσουμε κίνητρα για αύξηση των επενδύσεων. Ε, χρειαζόμαστε συνδεσιμότητα, αξιόπιστη. Δεν θέλουμε ένα νομοθετικό και γραφειοκρατικό τέρας. Θέλουμε επενδύσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις. Πρέπει, λοιπόν, να αναρωτηθούμε εάν επαρκεί το επενδυτικό μοντέλο που έχουμε αυτή τη στιγμή, αν χρειαζόμαστε διαφορετικό ή διαφορετικά πληθυντικό. Διασφάλιση επίση τη ουδετερότητα του διαδικτύου, αλλά για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να είμαστε γρήγοροι και αποτελεσματικοί. Και ε, κύριε Πρόεδρε, εδώ θα ήθελα να πω πως ε, υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ και κατά, αλλά όποιο επιθυμεί ε, υποδομέ που να που να βοηθούν χρειάζεται και προσπάθεια. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω πως ε, το σχέδιο έκθεσης ε, μπορεί να βελτιωθεί. Ε, σε γενικέ γραμμέ νομίζω πω έχει γίνει καλή δουλειά, όμω τα επιμέρου σημεία θα τα αναφέρω σε άλλη συζήτηση ή με τι ε, τροπολογίε μου. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρόιλ. Ο κύριο Χόκμαρκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την εισηγήτρια. Ήταν πολύ σύνθετο το καθήκον που ανέλαβα και ήταν εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. Τρία σημαντικά σημεία. Πρώτον, σε ό,τι φορά την ικανότητα, ε, πρέπει να είμαστε εδώ πιο ρεαλιστές. Εάν δεν έχουμε ε, αρκετά υψηλή ικανότητα, δεν ε, θα έχουμε καλά αποτελέσματα και θα δούμε νέο χάσμα στην Ευρώπη. Κάποιες χώρες θα κινούνται πιο γρήγορα, κάποιες λιγότερο και αυτό θα σημαίνει τεράστια προβλήματα για όλους μας. Ό,τι και αν πούμε για την ε, χωρητικότητα της τεχνολογίας, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει η ικανότητα και για τις οπτικές σύνες. Να τα δούμε τα υπόλοιπα, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί σε συγκεκριμένους στόχους. Τώρα, για τις επενδύσεις, νομίζω ότι θα δούμε πολύ διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό και για τις διάφορες ε, εξελίξεις των τομέα υποδομών. Είναι σημαντικό να υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Νομίζω ότι είναι καλό το όριο των 30 ετών, θα μπορούσαν και 25. Δεν πειράζει, αρκεί όμως να υπάρχουν κανόνες για την ανοιχτή πρόσβαση. Βλέπω ότι δεν έχω άλλο χρόνο. Εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία στην ε, εισηγήτρια. <laughs> Ευχαριστώ. πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω πως η έκθεση δείχνει πως το όραμά μας είναι καλύτερο από το όραμα της Κομισιόν και αυτή η έκθεση νομίζω μας δίνει την ευκαιρία να γίνει κάτι ουσιαστικό Εάν μάλιστα συνυπολογίσουμε και την ιδιότητα της ε, εισηγήτριας και των σχεδόν εισηγητών. Εάν δεν καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, τότε ε, θα επιδεινωθούν στο μέλλον. Το ζητούμενο εδώ είναι το φάσμα, το, 5G. Το 5G πρέπει να έχει εξαπλωθεί μέχρι το 2020. Υπάρχει μία ημερομηνία λοιπόν, αλλά ακόμα η Κομισιόν δεν έχει δώσει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Χρειάζεται λοιπόν αυτό να γίνει όχι σήμερα, χθε για να καταφέρουμε να φτάσουμε το 2020 και το 5G παντού. Η λύση πιστεύω δεν είναι ε, τίποτα άλλο από επενδύσεις, από κίνητρα. Ε, αυτή τη στιγμή οι επενδυτές δεν έχουν καμία διασφάλιση πως δεν θα ε, χάσουν τα λεφτά τους. Δεν υπάρχει σιγουριά. Χρειάζεται να διασφαλιστεί η συμβατότητα. Και αυτό αυτή τη στιγμή ακριβώς επειδή χαρακτηρίζεται από ασάφεια θα οδηγήσει σε χάος αν δεν ρυθμιστεί άμεσα. Δεν είναι μόνο βέβαια ευθύνη των εθνικών αρχών, αλλά πρέπει και εμείς να συνεισφέρουμε σε αυτό. Υπάρχουν ακόμα πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Γι' αυτό ελπίζω η συγκήτρια να καταφέρει να ε, επιλύσει αυτά τα προβλήματα. Λυπάμαι πολύ που δεν μπορώ να συνεχίσω, αλλά ένα λεπτό δεν φτάνει πραγματικά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Νομίζω πως πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταρχάς να οργανώσουμε οπτικές σύνες και 5G εδώ, μέσα στο κτίριο για να κάνουμε τη δουλειά μας. Πρώτα λοιπόν να δούμε αυτό. Επόμενος ο Αξελφός. Ευχαριστώ πολύ Πάουλ. Είμαι εισηγητή για το θέμα αυτό στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και αναρωτιέμαι ε, αν αυτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Καταρχάς ε, πρέπει να διερωτηθούμε πόσο ε, καινοτόμοι είμαστε και πόσο καινοτόμοι θέλουμε να γίνουμε. Και δεύτερον, τι ακριβώς θέλουμε από τις επικοινωνίες. Εάν υπό τις επικοινωνίες καταλαβαίνουμε και θέλουμε κάτι γενικό, τότε εντάξει, καλώς ήρθατε στο παρελθόν σας, διότι το χάσαμε το παιχνίδι. Υπάρχουν πολλά επίπεδα και δεν μπορούμε να τα υπολογίσουμε ούτε με αριθμούς, ούτε με διαφορετικούς τρόπους. Η επικοινωνία είναι καθημερινή, συνεχόμενη, από το αυτοκίνητο, στο δρόμο, ε, από το σπίτι, παντού. Γι' αυτό χρειάζεται να γίνει ένα τεράστιο άνοιγμα ε, στον ορισμό καταρχάς των επικοινωνιών. Τι είναι η επικοινωνία ε, και να συνδεθεί με την οδηγία για την ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο. Στο μέλλον πιστεύω δεν θα καταφέρουμε καμία πρόοδο εάν μένουμε στάσιμοι, εάν δεν αναγνωρίσουμε την ανάγκη για ουδετερότητα στην επικοινωνία, εάν δεν προσαρμοστούμε στις εξελίξεις. Ε, και αυτό λοιπόν χρειάζεται ριζική αναδιατύπωση του τι σημαίνει επικοινωνία. Δεν αρκεί ένα μοντέλο, δεν μπορούμε καν να δημιουργήσουμε ε, να επινοήσουμε ένα μοντέλο. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα μοντέλα είναι πολλά και να υπάρχει αυτή η δυνατότητα να αξιοποιηθούν. Γι' αυτό νομίζω πω σε συνδυασμό με όλα αυτά πρέπει να αναλύσουμε και να εξετάσουμε ταυτόχρονα την οδηγία για την ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φω. Ε, Κάποιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Βίλαν, εσεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την εξαιρετικά σημαντική συμβολή της ε, στη διαμόρφωση γνωμοδότη εδώ στο Κοινοβούλιο για την πρότασή μας. Βεβαίως ε, και χαιρετίζουμε την στήριξη της ε, σε μια σειρά στοιχείων της πρότασή μα και χαιρετίζουμε και το γενικότερο πνεύμα των παρεμβάσεων σήμερα το πρωί στην Επιτροπή για την ανάγκη υψηλού επίπεδου φιλοδοξίας σε ό,τι αφορά τα δίκτυα και την διασύνδεση στην Ευρώπη. Το να έχουμε λοιπόν όλα αυτά στην Ευρώπη θα είναι σημαντικό στόχος για μας. Θέλουμε κι εμείς και να σεβόμαστε τις αρχές της τεχνολογικής, τεχνολογικής ουδετερότητας, παράλληλα όμως να δίνουμε και κίνητρα ε, στις επενδύσεις, ιδίως ό,τι αφορά τις επενδύσεις υψηλού ρίσκου, που καλύπτουν πολλές ανάγκες και των ε, τελικών χρηστών στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στις επιχειρήσεις. Και αυτό αφορά και πολυεθνικές επιχειρήσεις ε, που πρέπει να χτίσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. Ε, είμαστε υπέρ και της φιλοδοξίας που σκιαγράφησε η συγγήτρια στην έκθεσή της ότι αφορά το ασύρματο δίκτυο. Νομίζω ότι πρόκειται για πολύ σημαντικό θεμέλιο της ανάπτυξης ε, της ε, νέας γενιάς ε, υπηρεσιών στην Ευρώπη, το 5G. Και χαιρετίζουμε και την έμφαση που δίνεται στις δοκιμασμένες αρχές της αγοράς. Νομίζουμε ότι όλα αυτά δίνουν ασφάλεια και προβλεψιμότητα στην αγορά, ενώ βέβαια απαιτούνται κοινέ προσπάθειες για να απλούστευθεί και να υπάρξει και σύγκληση στο κανονιστικό πλαίσιο σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πιλάρη Τεκαστήγιο, η συγγήτρια έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τις ε, παρεμβάσεις σας, για τις απόψεις σας. Ε, και ακριβώς ε, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε πρέπει να μοιραστούμε απόψεις, ε, να να συζητήσεις, να υποβληθούν οι τροπολογίες και να μοιραστούμε όλες αυτές τις ανησυχίες. Να συζητήσουμε και τα όσα δεν έχουμε ακόμα μέχρι σήμερα μπορέσει να συζητήσουμε. Γι' αυτό και είμαι απόλυτα ανοιχτή σε οποιαδήποτε, συζήτηση οποιασδήποτε πτυχής που περιλαμβάνεται εδώ, να συζητηθούν όλα ανοιχτά και βέβαια πολλά πράγματα θα αλλάξουν, είναι λογικό σε αυτή τη διαδικασία. Το σημαντικό είναι όμως να αλλάξουν προς το καλύτερο. Να έχουμε δηλαδή ένα σχέδιο το οποίο να είναι συνεπές και να βρει την στήριξη όλων. Γιατί αυτό είναι το κλειδί για να μπορέσουμε να έχουμε επιτυχία στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Πολύ το γνωρίζετε γιατί ε, έχετε συμμετέχει σε αντίστοιχες διαπραγματεύσεις. Τώρα έχουμε, τα διάφορα μοντέλα, ε, τη συν, ε, χρηματοδότηση, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να έχουμε μια πιο ευέλικτη δράση και να μιλήσουμε για εκείνες τις εμπορικές συμφωνίες που ενώ έχουν ε, χαρακτηριστικά παρόμοια ε, με τις ε, επενδύσεις να μπορούν να ληφθούν υπόψη. Και όχι να έχουμε μόνο την συν επένδυση, την κοινή επένδυση, που από την πλευρά της Κομισιόν φαινόταν να είναι το πιο αποκλειστικό. Τώρα όσον αφορά τα δίκτυα υψηλής ε, ταχύτητας και χωρητικότητας, ε, να πω δύο πράγματα. Ε, γιατί ακριβώς αυτό είναι το νομοθετικό πακέτο που πρέπει να συζητήσουμε και δεν θέλω να μακρηγορήσω. Τα, ο θέμα των δικτύων πολύ υψηλής ταχύτητας. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα, την Ισπανία, όπου ε, πραγματικά έχουμε φοβερή ταχύτητα. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια είμαστε στην πρωτοπορία. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη λοιπόν την ουδετερότητα των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται. Η ίνα αναφέρεται, αναφέρεται ο ορισμός και υπάρχει μια σαφής ένδειξη ότι αυτή είναι η τεχνολογία η οποία καλύτερα ανταποκρίνεται σε αυτούς τους στόχους της υψηλής ταχύτητας. Όμως θα πρέπει εδώ να συζητήσουμε για έναν ορισμό που θα καλύπτει και θα αγκαλιάζει τους στόχους που πρέπει να επιτυγχάνει οποιαδήποτε τεχνολογία εφαρμόζεται. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς ε, αυτά όλα θα ληφθούν υπόψη από, το εθνικό, από το εθνικό επίπεδο. Τα κράτη, οι εθνικές απαιτήσεις και η, τρόπος λειτουργίας είναι διαφορετικός πολύ και γι' αυτό και θα πρέπει να δώσουμε και κάποιο χώρο σε σχέση με το ποιες τεχνολογίες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν περισσότερο, περισσότερα πράγματα. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν. Και τέλος, σε σχέση με την επικοινωνία, τον... θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια, ένας γενικός ορισμός και υπάρχουν άλλοι που λένε ότι η ίδια η γενική έγκριση δεν είναι αμφισβητήσιμη. Πρέπει όντως να εφαρμοστεί. Αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να κάνουμε. Κατά τη γνώμη μου είναι μια σημαντική, μια καλή αρχή το να θέσουμε ήδη αυτήν την πρόταση της Κομισιόν, αλλά από εδώ και μπρος βέβαια μετά θα πρέπει να προσέξουμε ώστε να λάβουμε μια σωστή απόφαση. Το επιμένω, σημαντικό είναι να έχουμε μια στέρεη συμφωνία ε, για όλους που θα έχει μεγάλη στήριξη. Για να μπορέσουμε να ε, συμφωνήσουμε με όλα όσα επιθυμούμε και είμαι βεβαία ότι θα το καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια. Έχετε ένα δύσκολο έργο που πρέπει να ερμηνεύσετε τους νέους κανόνες, έχει αλλάξει και ο εσωτερικός κανονισμός τώρα και υπάρχει ο κανόνας 104. για αναδιατύπωση και, να, και θα ήθελα λοιπόν να σας ενημερώσω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 4η Απριλίου μέχρι τις 3 το απόγευμα. Όμως εδώ βλέπω ότι χρειάζεται και αιτιολόγηση των τροπολογιών. Αυτό το ξέρουμε και από τη διαδικασία του προϋπολογισμού, όπου πάντα μας ζητείται αιτιολογία για μια τροπολογία. Αυτά λοιπόν... Ε, Θέλω να σας πω, η γραμματεία θα σας στείλει και ένα email με τους ε, κανόνες, με όλες τις λεπτομέρειες του εσωτερικού κανονισμού που αφορούν αυτό το θέμα. Τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης για το Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Μπέρεκ. είναι ένα από τα θέματα τα οποία μας αφορά άμεσα και όλο ένα και αυξάνεται η σημασία του Μπέρεκ ακριβώς γιατί χρειαζόμαστε e ευφυή συστήματα τα οποία θα χειρίζονται την ψηφιακή αγορά. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο θέμα που έχει αρχίσει να συζητιέται, το μέλλον του Μπέρεκ και θα ήθελα να ανοίξει η συζήτηση δίνοντας το λόγο στον εισηγητή έτσι ώστε να μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσης. Έχετε τέσσερα λεπτά στη διάθεσή σας. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήδη αναφέρατε πολλά από αυτά που ήθελα να πω και εγώ. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω την σημερινή έκθεση το Μπέρεκ και η υπηρεσία Μπέρεκ είναι αποτέλεσμα ενός συμβιβασμού με το Συμβούλιο. Και αυτές οι διαπραγματεύσεις δεν ήταν καθόλου εύκολες. Από το 2009 και μετά νομίζω πως συγκεντρώσαμε αρκετή εμπειρία σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Μπέρεκ και αυτό που βλέπουμε είναι ότι όλα πάνε καλά. Το γραφείο Μπέρεκ, η επικουρική υπηρεσία και αυτή έχει δείξει πολύ καλή ε, λειτουργία. Σκοπός ε, είναι να αντλήσουν γνώση και από τα εθνικά δίκτυα και να γίνει σωστή ε, ανταλλαγή πληροφοριών. Μέχρι τώρα όλα ε, έβαιναν καλώς. Απλά τώρα υπάρχουν και πρόσθετες αρμοδιότητες για τον Μπέρεκ και το ερώτημα που έχουμε να απαντήσουμε είναι εάν αυτή η δομή που μέχρι τώρα λειτουργούσε πάρα πολύ καλά πρέπει να αλλάξει. Είμαι προσωπικά πεπισμένος ότι η ιδέα να συγχωνευτούν το Μπέρεκ και το γραφείο Μπέρεκ θα οδηγήσει σε τεράστιες επιπλοκές. Και θα γίνουν τα πράγματα πιο δύσκολα. Στην πρότασή μου που τροποποιεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν προτείνω να ακολουθήσουμε αυτή την πρόταση να παραμείνουν ανεξάρτητοι και ευέλικτοι αυτοί οι ε, φορείς ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών, διότι αυτό θα διασφαλίσει τον επαγγελματισμό και τη σταθερότητα γενικότερα. Ε, ας αφήσουμε τον ΠΕΡΕΚ να αναλάβει αυτές τις επιπλέον αρμοδιότητες, όμως ε, θα πρέπει να γίνει αυτό δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον. Και Είμαι επίσης πεπισμένος ότι το Μπέρεκ θα πρέπει να μείνει εκτός της άμεσης σφαίρας επιρροής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να μην διαταραχθεί η πολύ λεπτή θεσμική ισορροπία που με τόσο κόπο καταφέραμε να έχουμε. Φυσικά, πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και εκεί εστιάζει η έκθεσή μου. Προσπαθούμε να έχουμε μία καλή ε, αναλογία των θετικών στοιχείων από την εφιστάμενη δομή και των νέων προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω πως η πρόταση της Επιτροπής όντως είναι πολύ καλή σε ορισμένα σημεία. Για παράδειγμα, ε, σε ό,τι φορά τον Μπέρεκ υπάρχει ένα δίκτυο επικοινωνίας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν καλύφθηκε από τον κανονισμό του 2009. Μετά, το, συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο των ε, Ρυθμιστικών Φορέων του ΠΕΡΕΚ ε, έχει κάποια προβλήματα συντονισμού. Ε, ο διευθυντής τώρα του γραφείου ΠΕΡΕΚ προτείνω να κρατήσει το ρόλο που έχει και το Κοινοβούλιο επίσης να διατηρήσει την ε, παρουσαρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ταχθεί υπέρ της αποκέντρωσης των υπηρεσιών και με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Θα αυξηθούν οι απαιτήσει, γι' αυτό και προτείνω να αυξηθεί και το προσωπικό του Μπέρεκ. Και ε, αυτό ισχύει και για την ε, εσωτερική δομή του Μπέρεκ. Και επίσης πρέπει να ε, ενεργήσουμε έτσι ώστε να μην χρειάζεται να αλλάζει στο μέλλον κάθε λίγο η δομή του Μπέρεκ. Βλέπουμε πως ε, τα πράγματα εξελίσσονται, αλλάζουν. Πολλές φορές αναγκάζεται κάποιος να αναλάβει επιπρόσθετες αρμοδιότητες, γι' αυτό πρέπει ο κανονισμός να τροποποιηθεί καταλήλως. Ελπίζω με τους σκιώδες συζητητέ να έχουμε μια πάρα πολύ καλή έκθεση. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κάριντς έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Τοσνόσκι για το σχέδιο έκθεσης και για να συνοψίσω να πω πως οι γενικές γραμμές συμφωνώ με τις προτάσεις του. Εάν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια αγορά δημιουργώντας ε, μια υπηρεσία, τέλεια θα ήταν, υπέροχα. Ε, ενεργειακά, αν δούμε το θέμα, υπάρχουν, υπάρχει η αίσα, αλλά δεν υπάρχει ενιαία αγορά ηλεκτρισμού. Βλέπουμε τα προβλήματα, είναι μέρος του, της δέσμης μέτρων ε, που επεξεργαζόμαστε, αλλά το να δημιουργήσεις μια αγορά δεν σημαίνει απαραίτητο ότι πρέπει να δημιουργήσεις και μια υπηρεσία πιο πριν. Και το αντίστροφο, όταν δημιουργείς μια υπηρεσία δεν σημαίνει ότι μαζί της θα έρθει και μια νέα αγορά. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Στο ψηφιακό τομέα τώρα είναι αντίστοιχα τα πράγματα. Και πολλές φορές αυτό που δεν συνυπολογίζουμε είναι τα ε, ρυθμιστικά προβλήματα που αφορούν τον ανταγωνισμό, την έλλειψη ανταγωνισμού και τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Στην ουσία πρέπει να βρούμε τι δεν πάει καλά. Και όπως είπε και ο κύριος Στοσνόφσκι, ε, το ζητούμενο εδώ νομίζω είναι να ενισχύσουμε την υφιστάμενη δομή του Μπέρεκ χωρίς να ε, αλλάξουμε τίποτα στην ε, διοικητική του δομή στο οργανόγραμμα. Χρειάζεται δηλαδή το γραφείο Μπέρεκ ενίσχυση, προσωπικό, περισσότερα κονδύλια έτσι ώστε να η προσλάβει προσωπικό το οποίο θα αναλάβει αυτές τις ε, πρόσθετες ε, αρμοδιότητες. Συμφωνώ λοιπόν με τον κύριο Τσονόφσκι και όχι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο πολύ. Το θέμα δεν είναι να δημιουργήσουμε μία νέα υπηρεσία. Ίσως στο μέλλον να αποκτήσουμε περισσότερους λόγους για να το κάνουμε. Ε, θα έπρεπε αντίθετα να ενισχύσουμε τη λειτουργία των υφιστάμενων οργανισμών. Και να ενισχύσουμε λοιπόν την ε, περαιτέρω εξέλιξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Γι' αυτό θεωρώ πως σε αυτό το στάδιο καλύτερα είναι να αυξηθεί η χρηματοδότηση, να αυξηθούν οι αρμοδιότητες, αλλά να μην δημιουργήσουμε μία ε, επιπλέον δυσκολία, ανούσια δυσκολία με το να δημιουργήσουμε άλλη μία υπηρεσία. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σταματήσω εδώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή ε, με τον οποίο συμφωνούμε σε γενικές γραμμές. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κρέλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης. Εγώ θα δώσω μια διαφορετική κατεύθυνση στη συζήτηση. Η πολιτική μου ομάδα θεωρεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλή, σωστή και τη στηρίζει. Θεωρούμε πως είναι πολύ επίκαιρη σε μια εποχή που η ενιαία αγορά θέλει να ανοιχτεί στον τομέα των επικοινωνιών, χρειάζεται προσαρμογή, γι' αυτό θεωρώ πως ε, η η λειτουργία του Μπέρεκ και του γραφείου Μπέρεκ δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν αυτές τις ε, πρόσθετες αρμοδιότητες. Αν δούμε την δομή των οργανισμών αυτών ε, θα βρούμε πάρα πολλά, ε, πάρα πολλά προβλήματα, πολλή γραφειοκρατία. Και αν δούμε την πρόταση της Επιτροπής βλέπουμε πως μειώνεται η γραφειοκρατία με αυτό. Σίγουρα χρειάζεται να διασφαλιστεί η διαφάνεια, αλλά δεν μπορούμε να περιοριστούμε απλά δίνοντα ορισμένες συστάσεις. Υπήρξαν μάλιστα πολλές ε, περιπτώσεις ε, που ακριβώς λόγω της έλλειψης ε, εξουσίας για να προχωράει σε κάτι πέρα από συστάσεις, πολλές φορές ευχόμουν ο Μπέρεκ να είχε ήδη αυτές τις πρόσθετες αρμοδιότητες για να μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Νομίζω πως βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή που πρέπει να ληφθούν ορισμένες αποφάσεις. Ας μην βλέπουμε την Κομισιόν σαν τον εχθρό που βρίσκεται πάνω απ' όλα, πανταχού παρούσα και κάνει ό,τι θέλει. Ε, δεν δίνει η Κομισιόν ε, το βήμα για το τι θα κάνουμε. Νομίζω πως ε, πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που αλλάζει και για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την αλλαγή πρέπει να αναγνωρίσουμε τις νέες προκλήσεις και να τις δεχτούμε. Σίγουρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να μείνει εκτός. Σε αυτό είμαι 100% σύμφωνη. Πρέπει να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία των ε, οργανισμών. Γι' αυτό σε καμία περίπτωση δεν λέω κάτι το αντίθετο. Ε, και νομίζω πως παρά τις ε, διαφορές μας και τις διαφωνίες μας θα καταφέρουμε στο τέλος να συνεργαστούμε πολύ καλά και να δημιουργήσουμε ένα πολύ καλό σχέδιο έκθεσης. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κρέλ. Οι φιλελεύθεροι έχουν τώρα το λόγο. Κύριε Κάλλας. Ευχαριστώ πολύ. Κατανοώ το βασικό μήνυμα του εισηγήτου ότι δεν πρέπει να υπάρχει οργανισμός ή τόσο εκτεταμένος. Αλλά συμφωνώ και με τους προηγούμενους ομιλητές. Η ομάδα μου επίσης δεν θέλει τα χρήματα του Ευρωπαίου Φορολογούμενου ε, να πηγαίνουν ε, και να χρηματοδοτούν ένα απλό φόρουμ συζητήσεων. Έχω εξετάσει τις διάφορες ε, εκθέσεις για να κατανοήσω καλύτερα τα ζητήματα του κώδικα και σε όλες αυτές τις εκθέσεις ο Μπέρκ ουσιαστικά ζητάει εθνικές λύσεις. Πάντα βάσει δηλαδή, του εθνικού πλαισίου και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αυτό ισχύει στις περισσότερες των περιπτώσεων, όμως συμπεριλαμβάνει εκθέσεις και, και για τα OTTs και για τη διευκόλυνση του ίντερνετ των αντικειμένων όπου δεν μπορούμε να δούμε πώς γίνεται η εθνική αντιμετώπιση να είναι καλύτερη για τη δημιουργία οικονομίας κλίμακας. Επίσης, ό,τι φορά τις επιχειρήσεις ε, που ε, δραστηριοποιούνται διασυνοριακά, ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις B2B ε, λένε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ κρατών μελών, επομένω δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στο status quo αν θέλουμε μια καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία της ιστορικής αγοράς. Ναι, όντω δεν δημιουργείται έτσι μια νέα αγορά και εδώ συμφωνώ με τον κύριο Κάριντς, αλλά Ο σκοπό εδώ είναι η καλύτερη λειτουργία τη ενιαία αγορά. Ο Μπέρεκ πρέπει λοιπόν να διαματίζει καλύτερο, ε, πιο ενισχυμένο ρόλο για τι υπηρεσίε, το φάσμα, διασυνοριακέ υπηρεσίε και ομοιόμορφη ερμηνεία του ενωσιακού δικαίου. Πρέπει επίση ε, να ε, δώσουμε μεγάλη προσοχή στη διασύνδεση μεταξύ ε, του Μπέρεκ και του κώδικα, γιατί ο κώδικα αυξάνει την ευελιξία για τι εθνικέ ρυθμιστικέ αρχέ, να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό και να πετύχουν του στόχου συνδεσιμότητα. Όμω θα πρέπει να έχουμε κατά νου στην πρόταση αυτή και την καλύτερη διακυβέρνηση και έλεγχο του Μπέρεκ. Και έτσι για μα είναι πρόβλημα ω Άλντε να δώσουμε περισσότερο, μεγαλύτερο περιθώριο στι εθνικέ ρυθμιστικέ στι αρχές ε, να αυξήσουμε τις αρμοδιότητές του, αν δεν υπάρχει και ευρωπαϊκή εποπτεία. Και τέλος, ε, είναι ενισχυμένο ο ρόλο ε, τη Κομισιόν ε, στον ΜΠΕΡΕΚ. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είναι δορυφόρο ο ΜΠΕΡΕΚ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί η συνεργασία μεταξύ του ευρωπαϊκού και εθνικού πλαισίου είναι ουσιαστικά στοιχεία για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Πρέπει να υπάρχει μια δομή όμω που θα μα δίνει μια πραγματική ενωσιακή προσέγγιση σε ζητήματα που συνδέονται με την ενιαία αγορά και να μην έχουμε έναν απλό κοινό παρανομαστή ελάχιστο να να Ε, προσβλέπω στη συνέχιση των συζητήσεων και στη συνέχιση της συνεργασίας μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ράιμαν, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ τον εισηγητή για το προσχέδιο. Δεν θα πρέπει να βλέπουμε δύο πράγματα. Τις αρμοδιότητες και τη δομή του Μπέρικ δεν έχει νόημα για μένα να μιλήσω πρώτα για, το, για τη δομή και μετά να δούμε ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες στο μέλλον. Εάν δεν αλλάξουμε ε, τις αρμοδιότητες, εάν δεν διαβιβάσουμε πολύ περισσότερες αρμοδιότητες στον ε, ΒΕΡΕΚ, τότε δεν έχει τόση σημασία η δομή του. Εάν ε, προσθέσουμε πολλές αρμοδιότητες σε αυτόν τον οργανισμό, τότε βεβαίως χρειαζόμαστε έναν αυτόνομο, ανεξάρτητο, ε, ανεξάρτητο οργανισμό με εγγυημένη μάλιστα ανεξαρτησία και μετά πρέπει να δούμε και τους πόρους. Γιατί η ισχύ ε, του Μπέρεκ εξαρτάται και από τη χρηματοδότηση που θα πάρει. Και αυτό ισχύει για όλα τα κρατημέλη. Πρέπει να οργανώσουμε τον Μπέρεκ, ούτω ώστε και τα 28 κρατημέλη να δεσμεύονται να το χρηματοδοτήσουν. για να κάνει τη δουλειά του. Για μας λοιπόν είναι μια συνολική προσέγγιση. Εάν θέλουμε να φτιάξουμε έναν ισχυρό οργανισμό με πολλές αρμοδιότητες, ε, τότε ε, πρέπει να υπάρχει και ανάλογη στήριξη. Και εμείς ε, στηρίζουμε την ύπαρξη ενός ανεξάρτητου οργανισμού χωρίς επιρροές από τον, το πολιτικό στερεόμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρέιμον. Κύριος Μικ... Νίκα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να πω κάτι είναι θέμα αρχή καταρχάς. Είναι πολύ δύσκολο να ορίσουμε ποιο είναι ο ρόλος του Μπέρεκ στο μέλλον ακόμα και ε, ποιο είναι ο ρόλος των εθνικών αρχών. Ε, καταρχάς δεν θα πρέπει να έχουν καμία απολύτω σχέση με την πολιτική. Ούτε δηλαδή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως έχει προταθεί, ούτε και σε εθνικό επίπεδο δηλαδή, ούτε τα εθνικά κοινοβούλια. Και αυτό το λέω ακριβώς διότι πρόσφατα είδαμε με τα μάτια μας τι συμβαίνει όταν οι εθνικές αρχές ή γενικότερα οι αρχές αναλαμβάνουν αρμοδιότητες που ανήκουν στο Μπέρεκ. Για το 5G ας πούμε οι εθνικέ αρχέ δεν χρειάζεται να λάβουν καμία απόφαση, πρέπει απλά να εφαρμόσουν άλλε αποφάσει. Το μόνο που προσπαθούν να κάνουν είναι να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των ε, πελατών, των καταναλωτών. Και θα προσπαθήσω να σας ε, δώσω μία εικόνα το πώς βλέπω τα πράγματα. Ε, δεν μ' αρέσει η υπερβολική νομοθεσία και η ρύθμιση για το ένα, για το άλλο, για τα πάντα. Ξέρετε Μάλιστα ότι λέγεται και το ανέκδοτο ότι όταν οι δημόσιοι υπάλληλοι το πρωί ε, πίνουν τον καφέ τους και βαριούνται, δεν έχουν τι να κάνουν, λένε «Αχ, ας αποφασίσουμε να βασανίσουμε τον κόσμο, ας κάνουμε ένα νέο νομοσχέδιο». Ε, το Μπέρεκ λοιπόν πρέπει να βρει ένα όσο το δυνατόν βέλτιστο μοντέλο λειτουργίας και να επιλέξει από τις ε, καλύτερες πρακτικές των άλλων κρατών μελών. αναρωτιέμαι εάν κάτι που θα ε, αποφασιστεί, που αποφασίστηκε σε μία χώρα θα μπορεί να εφαρμοστεί σε μία άλλη. Δηλαδή γίνεται κάτι στη Ρουμανία, ας πούμε. Οι Γερμανοί θα το εφαρμόσουν. Έχουμε ε, πολλά κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει μία ανισορροπία δυνάμεων τι λέει το, τι άποψη έχει το Μπέρεκ, τι άποψη έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν υπάρχει κάποιο εδώ στην αίθουσα να μα πει, θα ήθελα πολύ να μάθω. Σα ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στον κύριο Βίζα Τυράβα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καθώς και την τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεση και την παρουσίαση των επιλογών που έχει ε, συστήσει στην Επιτροπή, που όπως θα έχετε παρατηρήσει διαφέρουν λίγο σε ορισμένες περιπτώσεις από τις δικές μας προτάσεις. Το πιο σημαντικό από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι έχουμε πάρει αυτή την διοργανική κοινή προσέγγιση για τους οργανισμούς ως ε, αφετηρία για τη συζήτηση αυτή με τους νομοθέτε. Βεβαίως είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε και ε, τις λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τον Μπέρεκ. Βέβαια, δεν είναι πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να ε, θίξει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία του Μπέρεκ ή των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Αυτό όμως που θεωρούμε σημαντικό, εφόσον υπάρχει και μια ευρεία συνένεση ότι θα υπάρξουν νέες σημαντικές αρμοδιότητες για τον Μπέρεκ, είναι να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα του Μπέρεκ. Υπάρχουν σήμερα σύνθετες δομές που μπορούν να απλουστευθούν. Η ανεξαρτησία των ε, εθνικών ρυθμιστικών αρχών και ε, η εμπειρογνωμοσύνη και δεξιότητες που παρέχουν αυτές οι αρχές θα είναι σημαντική πηγή για τον Μπέρεκ. Όμως πρέπει ε, να διαχειριστούν σημαντικοί πόροι απευθείας στον Μπέρεκ με μεγαλύτερη ευρωπαϊκή προσέγγιση σε σχέση με μια εθνική ρυθμιστική αρχή. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να έχουμε αυτή την ευρωπαϊκή προσέγγιση. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σιγητά, θα θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ όλους για αυτή την χρήσιμη συζήτηση. Αναμέναμε το μεγαλύτερο ζήτημα να είναι η απόφαση κατά πόσο πρέπει να αλλάξουμε την ε, οργανική σύσταση και θέση του Μπέρεκ. Ε, έχω πλήρη γνώση των νέων αρμοδιοτήτων που θα αναλάβει ο Μπέρεκ. Γι' αυτό και ήθελα το κείμενο να μείνει ανοιχτό, αν θέλετε, να μην ε, προσθέσω συγκεκριμένα όλες τις νέες αρμοδιότητες του Μπέρεκ. Ήθελα σκοπίμως να το αφήσω έτσι. Ευχαριστώ, λοιπόν, για τα όσα είπατε. Ήταν ακριβώς αυτό το πρόβλημα με το οποίο έχουμε έρθει να αντιμετωπί. Τώρα ένας οργανισμός δεν πρόκειται να ε, δημιουργήσει μια αγορά. Ήδη έχουμε 28 τέτοιους ε, οργανισμούς, τέτοιες αρχές. Παρ' όλα αυτά, όταν λαμβάνοντας υπόψη ε, και τη συμβολή των 28 Εθνικών Εθνικών Αρχών, έχει γίνει πλέον μια πολύ καλή δουλειά στον Μπέρεκ ε, υπάρχει πλέον ένα επαγγελματικό επίπεδο δράσης και θέλουμε να διατηρήσουμε αυτόν τον επαγγελματισμό και την ανεξαρτησία. Και να αποτελέσει και ένα φόρουμ όπου κάθε εθνική αρχή να μπορεί να εκφέρει γνώμη αναφέρθηκαν κάποια ζητήματα που μας δυσκολεύουν να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Όπως και να έχει, είναι μια ανοιχτή πρόταση αυτή που έχουμε υποβάλει. Είμαστε διεθυμένοι να εξετάσουμε κάποια από τα ζητήματα που θίξατε. Αλλά για να σχολιάσω αυτό που είπε η κυρία Κάλλας, δεν νομίζω ότι με το να δημιουργήσουμε έναν μεγάλο οργανισμό θα λύσουμε όλα τα προβλήματα. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα μας φέρει σε ακόμα μεγαλύτερες συζητήσεις στο Κοινοβούλιο για το αυξημένο κόστος και τα λοιπά. Έχω συζητήσει το θέμα της χρηματοδότησης με την Επιτροπή και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση και με τους σκιώδεις συζητητές. Προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας μας ε, και είμαι στη διάθεσή σας ε, για να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να διατηρηθεί και να μην ε, χάσουμε στην πορεία τον επαγγελματισμό και την καλή δουλειά που έχει κατακτήσει ε, ο Μπέρεκ, γιατί ε, την χάνει πλέον διεθνούς αναγνώρισης ο Μπέρεκ μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και έτσι και αυτό έχει μια αξία. Ακόμα και το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η γνώμη του Μπέρεκ όταν εξετάζουμε σύνθετα ζητήματα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Προθεσμή υποβολή τροπολογιών 30 Μαρτίου. Εξέταση τροπολογιών 11 Μαΐου. Ψηφοφορία στις 11 Ιουλίου 2017. Και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα αποφασιστεί στο μέλλον. Μετά περνάμε στην επόμενη έκθεση «Διαδικτυακή συνδεσιμότητα για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή. Ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit και του 5G». Η συγκητή είναι ο Μίχαλ Μπόνι από το ΕΛΚ και έχετε τέσσερα λεπτά καιρό για να κάνετε την παρουσίασή σας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις προτάσεις σας και τις ιδέες σας. Όσοι προλάβατε να στείλετε τροπολογίες, λάβαμε 250 τροπολογίες και πιστεύω πως το Κοινοβούλιο είναι ενωμένο και είχε την κοινή λογική να προτείνει συντονισμένα ένα σχέδιο δράσης για το 5G. Νομίζω πως σε γενικές γραμμές και η έκθεση και οι τροπολογίε ε, βρίσκονται στα ίδια με κυκλήματος. Μια που συζητάμε και για τον, ηλεκτρονικό, και τον, για τον ε, Ευρωπαϊκό Κώδικα Ελεκτρονικών Επικοινωνιών. Όπως ε, κατάλαβα υπάρχουν πέντε κύρια σημεία με τα οποία ασχολούνται οι τροπολογίε, ασχολούνται με την επιτυχία του δικτύου 5G, και αφορούν καταρχάς το ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο χρειάζεται απλοποίηση έτσι ώστε να είναι προσανατολισμένο στο μέλλον, να είναι υπέρ των επενδύσεων και υπέρ της καινοτομίας. Αυτό θα χρειαστεί μια αξιολόγηση ε, των ε, υποδομών για να δούμε αν ε, υποστηρίζουν τον ανταγωνισμό. Μετά χρειάζεται σαφής ορισμός ε, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δίκτυα υψηλής ικανότητας, όπως είπε και η κυρία Πιλάρτα Καστίγιο. Ε, δεν προτείνω την ύπαρξη αυτών των δικτύων στην έκθεση, όμως όταν θα έρθει η ώρα για να ε, προετοιμάσουμε τις τροπολογίες θα το προσθέσω. Έπειτα, χρειάζεται ένα σαφές πλαίσιο για την ανάπτυξη των επενδύσεων. Χρειάζεται οι επενδύσεις να έχουν απόδοση, όμως για να γίνει αυτό πρέπει να διασφαλιστεί ασφάλεια και ε, ο μακροπρόθεσμος χαρακτήρας τους. Γι' αυτό λοιπόν ε, ε, στο θέμα των αδειών μπορούμε να εξετάσουμε αυτές τις επιτυχίες. Ξέρω πως ορισμένοι συνάδελφοι είναι υπέρ των μακρο... μακροχρόνιων αδειών. Μετά, εναρμόνιση το δίκτυο 5G απαιτεί εναρμόνιση των αποφάσεων που αφορούν το ραδιοφάσμα. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος ε, για καθυστερήσεις και θα έπρεπε να υπάρχει αναγκαία ευελιξία έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να σχεδιάσει το δικό του δίκτυο εφόσον βέβαια υπάρχει και η δυνατότητα και να επιλέξει από 2G, 3G, 5G, δορυφορική επικοινωνία κτλ. Και καθώς και να συνδέσει όλα αυτά. Χρειάζεται, χρειάζονται οι συχνότητες 26 και 28 GHz, α, καθώς, και, ε, καθώς γιατί υπάρχουν πολλές χώρες που, ε, όπως η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, ε, που... Ε, ανταγωνίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, η διαχείριση του ραδιοφάσματος θα πρέπει, πιστεύουμε, να αναλυφθεί από τον Μπέρεκ, χωρίς ακόμα να ξέρουμε όμως τι ακριβώς θα κάνει. Πρέπει να καταλάβουμε πως ο Μπέρεκ δεν είναι ένας ακόμα από, από τους πολλούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Ε, αν εναρμονίσουμε την νομοθεσία για το ραδιοφάσμα, θα έχουμε ε, την ε, δυνατότητα να πετύχουμε και τους άλλους στόχους. Αν δεν το κάνουμε δεν μπορούμε και εδώ μπορεί να παίξει ε, το ρόλο του ο και Επίσης, ας αναλογιστούμε και το κόστος εφαρμογής του 5G και το τι μπορεί να σημαίνει καθυστέρηση της εφαρμογής του, στην εφαρμογή του 5G για την οικονομία μας. Είναι πολύ σημαντικό Εκεί λοιπόν αυτή η ρυθμιστική επικαιροποίηση. Μετά, για να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό, ε, χρειάζεται δράση. Υπάρχουν διάφορες πτυχές του κατακαιρματισμού, υπάρχει ο διαχωρισμός ανάμεσα σε αστικά κέντρα και ε, ύπεθρο, σε ε, διανομή συχνοτήτων του φάσματος και μετά και ένας οδικός χάρτης, ο οποίος χρειάζεται σαφές χρονοδιάγραμμα και η βιομηχανία επίσης πρέπει να παίξει το ρόλο της. Αυτή τη στιγμή, χωρίς τη συμμετοχή όλων αυτών, δεν μπορούμε να έχουμε επιτυχία στο, στο, στο να δημιουργήσουμε το 5G. Χρειάζεται λοιπόν ένας οδικός χάρτης ε, που θα αναφέρεται στη χρηματοδότηση των επενδύσεων και ελπίζω να καταφέρουμε με τους κοιότητες εισηγητές να συντονιστούμε έτσι ώστε να δώσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα κράτη-μέλη αλλά και σε όλους τους ε, ενδιαφερόμενους φορείς ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το χρηγορότερο δυνατόν η και εμ, καθολική εφαρμογή του 5G. Στις 25 Απριλίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Ήτρε τη ε, συμβιβαστικές τροπολογίες γενικότερα τη τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Βέρνερ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον, πρόεδρο, τον ε, εισηγητή κύριο Μπόνι για την πολύ καλή δουλειά που έκανε είναι ένα τεράστια σημασία θέμα. Έχουμε και την πρόταση από τον περασμένο Σεπτέμβριο και πρέπει επιτέλους να επιταχύνουμε τα πράγματα έτσι ώστε να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Αυτή τη βδομάδα στην έκθεση ΣΥΜΠΙΤΕ στο Ανόβερο η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι όλα τα δημόσια κτίρια, σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες και τα λοιπά, ιδιαίτερα όσα βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, θα πάρουν ε, κουπόνια, ας πούμε, πιστώσεις ε, για να αποκτήσουν ε, πιο γρήγορα από τους άλλους ε, πρόσβαση στο δίκτυο 5G και, στα, και στα, σε ταχύτητα gigabit. Αυτό πιστεύω πως είναι ενδεικτικό του τι μπορούμε να κάνουμε. Νομίζω πως υπάρχει καλή ε, συνέργεια ανάμεσα σε όλους τους φορείς και θα ήθελα να σταθώ σε πέντε, ε, πέντε περίπου σημεία. Καταρχά πρέπει να σκεφτούμε συνολικά τα πράγματα και τον καταναλωτή και το δίκτυο και την ταχύτητα και να δούμε ότι θα καταφέρουμε να φτάσουμε το στόχο του 5G μόνο όταν υπάρχει η κατάλληλη, το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο και χωρί να ξεχνάμε ποτέ ότι ο καταναλωτή ε, βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντό μα. Μετά, ανεξάρτητα από μια ανεξάρτητη δυνατή υποδομή, χρειάζεται μία ε, εστίαση στις ε, ιαλοίνες. Αυτές οι οπτικές ίνες είναι ε, απαραίτητες σχεδόν για την εξάπλωση του 5G. Μετά, χρειάζεται μεγάλο ποσοστό κρατικών επιχορηγήσεων βέβαια, αλλά νομίζω πως η πλειοψηφία της χρηματοδότησης θα προέλθει από τον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό Πρέπει να αναγνωρίσουμε ε, το πόσο σημαντικό είναι να δοθούν κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα, γιατί μπορεί να επηρεάσει άμεσα και κάθετα τις εξελίξεις. Τέταρτον, έτσι ώστε να τονωθεί η οικονομία, να τονωθεί η καινοτομία, οι επενδύσεις πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει το δίκτυο 5G μέχρι το τέλος του χρόνου. Ανεξάρτητα αν αυτό θα γίνει πρώτα στις πόλεις, θα γίνει στην Ήπεθρο κτλ. Αυτά λοιπόν τα ολίγα από εμένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά τον κύριο Μπόνη και, ε, να, και θα χαρώ πολύ για, για τη συνεργασία με τους υπόλοιπους και οδησυχητές. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τοσενόφσκι έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ. Ε, τη απουσία του σκιαδησηγητή τον αντικαθιστώ. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την εκτίμησή μου για την προσέγγιση του εισηγητή. Η έκθεση αυτή είναι τμήμα του ισδέσμες για τις τηλεπικοινωνίες και η δέσμη αυτή δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη. Η έκθεση λοιπόν αυτή εστιάζει ιδιαίτερα στο μέλλον Εμεί δηλαδή φτιάχνουμε κανόνε που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται στο μέλλον και ήθελα λοιπόν να εκτιμήσω και να, να εκφράσω την εκτιμήσή μου και να στηρίξω το όσα είπε ο εισηγητή, ότι δηλαδή πρέπει να βρούμε απλού κανόνε να μην κάνουμε ένα περίπλοκο ρυθμιστικό πλαίσιο εξ αρχή. Βέβαια αυτό θα οδηγήσει και στην προσέλκυση επενδύσεων στα δίκτυα 5G που θα αντιπροσωπεύουν ένα τελείως νέο τεχνολογικό βήμα ε, συμφωνώ με τον εισηγητή ότι το περιβάλλον θα πρέπει να είναι προβλέψιμο και σε ξεκάθαρο για τους επενδυτές. Συμφωνώ επίσης με το όσα είπε για τις ε, προσδοκίες του Μπάρακ. Έχουν εμπειρία από τις δυσκολίες του παρελθόντος και έτσι θα μας βοηθήσουν να προετοιμάσουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι καθοριστική σημασία για την γρήγορη ε, ανάπτυξη του 5G. Σας ευχαριστώ πολύ και συμφωνώ και με την προσέγγιση της, ε, του εισηγητή στην έκθεση. Ε, είναι, όπως είπαμε, αναπόσπαστο στο τμήμα της δέσμης που θα συζητηθεί φέτος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πλάνκο Λόπεθ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εν γέννη, συμμερίζομαι την άποψη της Κομισιόν σε σχέση με την κοινωνία των Gigabit. Ωστόσο, Πιστεύω πως για να το καταφέρουμε αυτό θα είναι σημαντικό να αποφύγουμε την έλλειψη συντονισμού όπως ε, που, είχαμε με το 4G που μας οδήγησε σε σημαντική καθυστέρηση. 86% κάλυψη. Έχουμε και μόνο 36% ε, ε, στις χορτικές περιοχές. Γι' αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε προς μια κοινωνία ε, ένταξης όπου θα υπάρχει πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες σε όλη την επικράτη της Ένωσης και σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Επίσης πιστεύω ότι σε όλα αυτά σε ρόλο κλειδί παίζει η επένδυση στην παιδεία ώστε να μορφωθούν πολίτες που θα είναι ικανοί να χειριστούν διαχειριστούν τις ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά και να καταλάβουν τις επιπτώσεις τους στην άσκηση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και άρα για να έχουν πολύ υψηλέ ε, δεξιότητες όταν και προσόντα όταν θα πρέπει να μπουν στην αγορά εργασίας. Σα ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Πιλάρντε Καστίγιο. Ένα λεπτό για να εκμεταλλευτώ και την ε, παρέμβαση του συναδέλφου Μπόνι για να υπογραμμίσω μια πτυχή του φάσματος. Ε, επέμεινε και είναι όντως πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη των δικτύων 5G. Εγώ ε, το κάνω και το ίδιο, το είπα και πριν, αλλά πρέπει να αναφέρω και πάλι ένα θέμα συγκεκριμένο, την διάρκεια της άδειας, της αδειοδότησης. Δεν υπάρχει περίπτωση μια μεγάλη επένδυση να μην συνοδεύεται από μια αδειοδότηση για, μια μεγάλη, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εκμετάλλευσης της εν λόγω επένδυσης. 56 GHz σημαίνει φάσμα επιπλέον και αυτό σημαίνει μεγάλες επενδύσεις. Ε, το Κοινοβούλιο μονίμως και σταθερά έχει στηρίξει τη διεύρυνση της, την, την παράταση της ισχύουσας διάρκειας. 25, 30, 25 χρόνια, όπως ε, προτείναμε και εγκρίναμε στην νέα χώρα για τις τηλεπικοινωνίες. Πάντως, οι αναλυτές των επενδύσεων ακριβώς λένε ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η συσχέτιση ανάμεσα στις επενδύσεις και τους όρους ε, εκμετάλλευσης και υπογράμμιζαν ότι σε, στις περιπτώσεις, σε θέματα μαλλοφάσματος η άδεια εκμετάλλευση θα πρέπει να είναι μακρόχρονη. Και υπάρχουν και μηχανισμοί για να ελέγξουμε ότι αν δεν υπάρχει αρκετή χρήση του φάσματος μπορεί και να το χάσει η ο δίουχος. Αλλά πάντως είναι απαραίτητο και ζητώ από όσους θα ασχοληθούν με αυτό το θέμα και έχουν ευθύνη ε, για αυτό το φάκελο να, προσεγγίσουμε, να το προσεγγίσουμε με αυτή την αντικειμενικότητα ε, για να μπορέσουμε έτσι να προωθήσουμε τις επενδύσεις σε αυτό το ε, τομέα. Κομπούλα νάτρι τώρα. Ναι, για το φάσμα πρέπει πολύ προσεκτικά να δουλέψουμε, αλλά πάνε χέρι-χέρι. Και ε, ο εισηγητής αφαίρεσε την ανάγκη για μοιρασιά. Υπάρχει νέα ανάγκη λόγω του 5G. Επίσης, αν δεν το χρησιμοποιείς θα το χάσεις αυτή η αρχή. Αλλά και πάλι θα πρέπει να δούμε τι ισχύει για τον αδιούχο εκμετάλλευσης. Ε, γιατί όλα αυτά θα πρέπει να συμβαδίζουν. Λυπούμε και πάλι που σας λέω, αλλά το 5G δεν είναι μόνο η επικοινωνία, μόνο δεν είναι μόνο οι υπάρχοντες φορείς που θα το χρησιμοποιήσουν. Θα είναι και νέοι φορείς στην αγορά και θα ήθελαν να είναι Ευρωπαίοι θα, θα ήθελα η ψηφιοποίηση να ωφελήσει την Ευρώπη. Όχι η Ασία να βιάχνει τον εξοπλισμό και η Αμερική το περιεχόμενο. Πρέπει να έχουμε αυτή την προστέμενη αξία για την Ευρώπη. Τώρα δεν υπάρχουν πρότυπα για το 5G ακόμα και δεν μπορούμε να αποφασίσουμε. Αλλά από όσα άκουσα δεν αρκεί οι, οι κινητές ε, κεραίες. Χρειάζεται και μια ραχοκοκαλιά. Και όπως είπε και ο Μάρτιν, αυτό είναι οι Ίνες. Είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανεί ότι χάλκινα καλώδια θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά για το 5G. Και αυτό πρέπει να το αναφέρουμε. Πρέπει να είμαστε ουδέτεροι τεχνολογικά, με την έννοια ότι η ραχοκοκαλιά πρέπει να είναι σε κάθε χώρα και σε κάθε σημαντικό. Διάβασα τα νέα ε, ότι εγκρίθηκε 48 γίγα αναδευτερόλεπτο ε, εγκρίθηκε η μεταφορά δεδομένων μέσω του φωτός. Μέχρι ότου αυτό να μπει σε εφαρμογή όμως, πάλι χρειαζόμαστε τις σύνες. Το 5G είναι μελλοντική τεχνολογία, δεν μπορούν να γίνουν όλα με βάση την παλιά τεχνολογία. Αυτό πρέπει να πούμε στους επενδυτές είναι να μην επενδύσουν περισσότερο σε κάτι το οποίο είναι στη λήξη του. κύριος Έριξον ε, είναι υπουργό στην Σουηδία τώρα και φτιάχνουν τώρα τα σπίτια ένα, για ένα γίγα. Ναι, στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι διαφορετικέ οι ανάγκε, αλλά πρέπει εμεί να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ετοιμαστούν όλα τα κρατημέλη για το 5G. Ο κύριος Ζαχίνιο ε, τώρα παρακαλώ. Να, συγγνώμη, δεν φορούσα το, τα ακουστικά μου. Σα ευχαριστώ πολύ. Εγώ ήθελα να χαιρετήσω την εργασία, την εξαιρετική εργασία του εισηγητή και να υπογραμμίσω την ολοκληρωμένη προοπτική με την οποία εκπονήθηκε αυτή η έκθεση, παράλληλα με άλλες εκθέσεις ε, που καλύπτουν τις διάφορες διαστάσεις της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής κοινωνίας των γιγαμπίτ. Ε, ε, οι προτάσεις ε, θα αξιολογούνται και προσπάθησα να δώσω μεγαλύτερη έμφαση σε δύο θέματα που είναι πολύ σημαντικά κατά τη γνώμη μου. Πρώτον, η καθολικότητα είναι, για, είναι η πολύ σημαντική. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια διπλή, ένα διπλό αποκλεισμό για τους πολίτες. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλη τη δυνατότητα, όλες τις δυνατότητες που έχουμε, ώστε να είναι καθολική αυτή η δυνατότητα ε, και να τονίσουμε την ποιότητα της εμπειρίας. Ναι, το ίντερνετ πρέπει να είναι ουδέτερο, οικονομικά θα πρέπει να εγγυηθούμε τη μεγαλύτερη δυνατή ουδετερότητα, όμως η ποιότητα θα πρέπει αυτή να προστατευτεί. Να τονίσω επίσης ότι η πρωτοβουλία Wi-Fi for You θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να λυθούν κάποια από αυτά τα ζητήματα. Με αυτή την πρωτοβουλία έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο πιλωτικό πρόγραμμα που να αποτελεί μια οπτική αναφορά, να δείξει στους Ευρωπαίους και στον κόσμο γιατί είχαμε και τη συζήτηση για τις ε, ψηφιακές πλατφόρμες, να δείξει λοιπόν ποια είναι η ευρωπαϊκή, το ευρωπαϊκό όραμα για την ανάπτυξη της νέας ψηφιακής κοινωνίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή κύριο Μπόνι για αυτό το σχέδιο έκθεσης. Το σχέδιο έκθεσης είναι αρκετά επίκαιρο δεδομένη της ταυτόχρονης ψηφοφορίας τώρα ε, σε Επιτροπή και πιστεύω πως θα στείλει ένα σαφές μήνυμα όχι μόνο για το νομοθετικό έργο που γίνεται στην Επιτροπή, αλλά και για ένα εύρος άλλων δραστηριοτήτων που γίνονται αυτή τη στιγμή χωρίς ε, τη διαδικασία της, ε, των συνομοθετών για το ραδιοφάσμα ή ε, επίσης γίνονται και πολλά σε εθνικό επίπεδο που στόχο έχουν στην ανάπτυξη αυτού του δικτύου, τη συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους φορείς και στην αγορά και αυτής της ε, κάθετη οικονομία, όπως ε, λέμε. Σημαντικό είναι να δώσουμε την κατάλληλη δομή, μια αρκετά φιλόδοξη δομή, έτσι ώστε να μπορούμε να τα επεξέλθουμε στις ανάγκες που θα υπάρχουν μέχρι το 2025 όπου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβεί σε μια νέα εκτίμηση του τι χρειάζεται. Τόσο για τον τομέα των επιχειρήσεων, όσο για τους ιδιώτες, τους πολίτες και την εκπαίδευση. Λοιπόν, είναι μακροπρόθεσμο το όραμά μας, γι' αυτό χρειάζεται μια πολύ συγκεκριμένη εντελεχής αξιολόγηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ο λόγος πίσω στον εισηγητή, κύριο Μπόνη. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις προτάσεις σας. Έχω αναλύσει όλες τις τροπολογίες και νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι αυτή η έκθεση θα προηγηθεί της νομοθεσίας. Επομένως μπορούμε να την αξιοποιήσουμε ως ένα μέσο προώθησης ε, του 5G. Και όπως αναφέρθηκε είναι σημαντικά τα όσα συμβαίνουν στη Γερμανία και τα όσα θα υπογραφούν αύριο στη Ρώμη ε, με τους εκπροσώπους όλων των ευρωπαϊκών χωρών και την κοινή τους ε, δήλωση για τα αυτοματοποιημένα οχήματα. Επομένως, είναι σημαντικό να διαμορφώσουμε ένα υπόβαθρο κοινή ε, αντίληψης για το 5G, γιατί στη συνέχεια θα είναι πιο εύκολο να εργαστούμε για το μέλλον, να υλοποιήσουμε την ε, νομοθεσία μας και να έχουμε έτσι ένα θετικό ε, κλίμα και στις σχέσεις μας με τους ε, καταναλωτές. Γιατί και αυτοί πρέπει να κατανοήσουν όλες τις νέες ε, ευκαιρίες που θα τους παρέχει το 5G. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Θα εργαστούμε επί των συμβαστικών τροπολογιών και ελπίζω εγκαίρως να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπόνη. 25 Απριλίου λοιπόν θα γίνει η ψηφορία στην Ήτρε και μάλλον τον Ιούνιο στην Ολομέλεια. Φτάνουμε τώρα στο τελευταίο σημείο της μέσης διάταξης τώρα, αποστολή της Επιτροπής Ήτρε στο 11ο συνέδριο του Φόρουμ για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου IGF στο Μεξικό η κυρία Δελκαστήλιο να μας ενημερώσει για δύο λεπτά για τα όσα συνέβησαν ε, στο Μεξικό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, πολύ σύντομα γιατί υπάρχει μια πάρα πολύ καλή έκθεση την οποία μπορούν να διαβάσουν όλα τα μέλη. Και εκεί παρουσιάζονται όλα λεπτομερέστατα. Να πω μόνο ότι ήταν η ενδέκατη συνεδρίαση του, ε, του φόρουμ, το ενδέκατο συνέδριο του φόρουμ για τη διακυβέρνηση. Θέλουμε να ε, αυξήσουμε τι δυνατότητε για ένα συμπεριληπτικό διάλογο και την, ε, για, για τα ζητήματα διακυβέρνηση, να δώσουμε τις ευκαιρίες εντοπισμού των βέλτιστων πρακτικών και να τα επισημάνουμε όλα αυτά στους αρμόδιους φορείς αλλά και στην κοινή γνώμη. Όλα αυτά για να ενισχύσουμε την οικοδόμηση δυναμικού στην διακυβέρνηση διαδικτύου. Είχαμε μια αρκετά μεγάλη ε, αντιπροσωπή από επιμέρους επιτροπές, 11 μέλη συνολικά, που εκπροσωπούσαν διάφορες ε, επιτροπές. Και πάλι φάνηκε ξεκάθαρα πόσο σημαντικό είναι να έχουμε αυτό το βήμα, αυτή την πλατφόρμα, για να εντοπίσουμε, όπως είπα και προηγουμένως, ε, τέτοια ζητήματα που ανακύπτουν, να ανταλλάξουμε απόψεις, ε, να γίνει αυτός ο διάλογος ήταν και πάλι τόσο ξεκάθαρα. Από πρακτικής άποψης είχαμε διάφορες ε, συνεδριάσεις με ενδιαφέρονους φορείς, ε, με εκπροσώπηση της Google, Ένωση Προοδευτικών Τηλεπικοινωνιών, από τον ακαδημαϊκό χώρο, από οργανώσεις προστασίας ανηλίκων, Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή σε μία πλειάδα σεμιναρίων και συνεδριάσεων. Εγώ συμπεραίνω ότι ως Κοινοβούλιο, ως Επιτροπή Ήτρε, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από πλευρά τη, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί έχουμε ισχυρή παρουσία σε αυτή την πλατφόρμα Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν, αλλά και εμείς ως Κοινοβούλιο. Νομίζω λοιπόν, κλείνοντας, ότι πρέπει να επιδιώξουμε την ε, διατήρηση αυτής της πλατφόρμας με τη σημερινή της μορφή, γιατί όλο ένα και ενισχύεται ο ρόλος μας εκεί και καλό και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, ξεκινώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να αυξήσουν τη δύναμή μας ε, και την παρουσία μας εκεί. Ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν βλέπω να έχει ζητήσει κάποιο άλλο το λόγο για αυτό το θέμα. Εδώ λοιπόν ολοκληρώσαμε την πρωινή μας συνεδρίαση και θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή ότι σήμερα θα συζητήσουμε το ενεργειακό πακέτο με μια κρόαση στις 3 το μεσημέρι. Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους λοιπόν και σας καλώ όλους να είστε εδώ. Τέλος της συνεδρίασης.